Καθίστε παρακαλώ. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Γεωργία η σημερινή αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο είναι πολύ μεγάλη χαρά μου. Καλωσορίζω τον Επίτροπο Τσιόλος εδώ. Θα περάσουμε το απόγευμα μαζί να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η παρουσία του Επιτρόπου ΔΕ δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσουν τα θεσμικά όργανα και ότι είναι ενωμένα είναι σαφής λοιπόν η συνεργασία μας και σε θεσμικό επίπεδο. Η συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν σίγουρα έχει διευρυμένες εξουσίες με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνα στο Κοινοβούλιο για να, να βαθμιστεί το δημοκρατικό προφίλ τη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μας τον ε, Επίτροπο είναι στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ο Επίτροπος ε, Ημικύκλιο για πρώτη φορά. Και πραγματικά αυτό αποδεικνύει και τη δέσμευσή σας για συνεργασία με την Επιτροπή μας. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει ξεκάθαρα τη σημασία που αποδίδουν οι Ευρωπαίοι πολίτε σε αυτόν τον τομέα. Είναι μια μεγάλη μέρα, είναι ακόμη ένα σημαντικό βήμα προ τη μεταρρύθμιση μια άκρο σημαντική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. την πλέον σημαντική πολιτική πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός και για την ανάπτυξη του ήθους και του πνεύματος ε, του κοινοτικού. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Το ψήφισμα της 8 Ιουλίου για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής μέχρι το 2013 ήταν η αρχή. Και σήμερα έχουμε το αποκορύφωμα, το επιστέγασμα αυτής της διαδικασίας. Ο Επίτροπος θα μας μιλήσει για κάποιες από τις επιλογές και τις ε, αποφάσεις που ελήφθησαν. Πριν του δώσω το λόγο θέλω να επαναλάβω τη μεγάλη σημασία της σημερινή εκδήλωσης. Είμαστε εδώ όλοι μαζί, εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε για να εγκρίνουμε τα επόμενα μέτρα τα οποία θα φέρουν σε αισιοπέρα στην μεταρρύθμιση. Είχαμε αποκλίνουσες απόψεις, ίσως και έχουμε αποκλίνουσες απόψεις, αλλά αυτό είναι ο πλούτος που μπορούμε να συνεισφέρουμε στη συζήτηση. ώστε να εξελιχθεί ο τομέας της γεωργίας, να αναπτυχθούν ε, τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ σήμερα ιδίω όσου έρχεστε για πρώτη φορά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε μάλιστα μέχρι και από τι Αζόρε προσκεκλημένους. Ε, θέλω να σα καλωσορίσω όλου, να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα και να δώσω χωρί χρονοτριβή το λόγο στον Επίτροπο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Θα ήθελα ε, πρώτα απ' όλα να εγγράψω τη σημερινή μας συζήτηση σε ένα θα έλεγα πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο. Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον ε, μιας κρίσιμη επιλογής για μια ολόκληρη γενιά. Δηλαδή, επιλογή ανάμεσα σε μια ε, γεωργία που θα καλύψει όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια ή μια γεωργία που θα περιθωριοποιηθεί ε, ε, οικονομικός πώς και κοινωνικός πώς. Είναι μια οικονομική επιλογή και επιλογή τρόπου ζωής για την ποικιλότητα, για την αυθεντικότητα, για την ποιότητα, για τις βασικές αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού ή μια επιλογή σχετικά με το πώς το ιδανικό μας ε, θα μπορούσε να επιβιώσει σε μια ενωμένη και Ευρώπη και θα δούμε με ποιους τρόπους μπορεί να συμβεί αυτό, ποια θα είναι η έκφανση αυτού του ιδανικού μέσα στην κοινωνία μας. Ε, Ορισμένες φορές ε, καλούμαστε να κάνουμε ψευδείς επιλογέ ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, Φερρυπίν. Εγώ θα σας προτείνω σήμερα ένα όραμα που αντιβαίνει σε αυτό το ψευδοδήλημα διότι είμαι πεπισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε διάφορα επίπεδα, από το παγκόσμιο μέχρι το τοπικό, ε, λαμβάνοντας, εξακολουθώντας να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες της κοινωνίας μας και καλύπτοντας τις βαθύτερες ανησυχίες της κοινωνίας μας. Ε, ε, τα εργαλεία της κοινή γεωργικής πολιτικής έχουν κέρια σημασία για να ε, επιτευχθούν οι στόχοι της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020. Επίσης, η κοινή γεωργική πολιτική μπορεί να αποτελέσει αγαστό παράδειγμα σχετικά με το πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την βιωσιμότητα ή τις οικονομικές μας επιδόσεις. Η ανακοίνωση που εισηγούμε σήμερα ε, οδηγεί σε ένα άνοιγμα τη κοινή γεωργική πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τι σημερινέ προκλήσει, ε, διατηρώντα τον κεντρικό ρόλο βέβαια τη γεωργία, ε, δηλαδή παραγωγή τροφίμων. Ο στόχος είναι στην καρδιά της κοινή γεωργικής πολιτικής, μία κοινή γεωργικής πολιτικής που σήμερα είναι προσανατολισμένη στην παραγωγή τροφίμων. Η καρδιά λοιπόν της κοινή γεωργικής πολιτικής να συμπεριλάβει και άλλα στοιχεία όπως διαχείριση φυσικών πόρων, ε, επίτευξη ε, ισορροπίας ε, ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό το διευρυμένο πυρήνα μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερες προσδοκίες της κοινωνίας ε, και να η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική θα λαμβάνει διόντως υπόψη περισσότερο εν πάση περιπτώσει σε σχέση με σήμερα ε, την ανάγκη της ε, βιοπικιλότητας. Αυτός ο στόχος καλύπτει ολόκληρη την κοινωνία και οι πόροι θα... Υπάρχουν πάρα πολλοί πόροι που είναι στη διάθεση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Επανειλημμένα έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα θα επανέλθω στη συνέχεια, αλλά θα ήθελα πρώτα να ξεκαθαρίσω με ποιο τρόπο η κοινή γεωργική πολιτική, όπως στηρίζεται από ολόκληρη την κοινωνία, θα ε, βρεθεί στη θέση να ανταπεξέλθει στις ε, νέε προκλήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινεί. Ε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική σήμερα διέρχεται μια κρίση νομιμότητας περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό δεν είναι νέο στοιχείο δεν είναι στοιχείο των τελευταίων μηνών, δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Η καλύτερη στρατηγική για να διατηρήσουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε για την κοινή γεωργική πολιτική είναι να ανοίξουμε αυτή την κοινή γεωργική πολιτική ούτως ώστε να ε, καλύψει ε, τις ανησυχίες ε, ευρύτερων πληθυσμιακών ομάδων της κοινωνίας μας σε σχέση με τις ανησυχίες κάποιων ε, και πιο συγκεκριμένα των γεωργών, θα ήθελα να ερμηνεύσετε αυτά που λέω στο πλαίσιο της ε, επιδίωξη τη νομιμοποίηση κοινή γεωργική πολιτική, ώστε να καλύψει τι προσδοκίε των πολιτών. Νομίζω ότι είναι η σωστή στιγμή τώρα για να προβούμε ε, σε μεταρρύθμιση. Δεν είναι αργά, δεν είναι νωρί, είναι ακριβώ η κατάλληλη στιγμή. Οι αγρονομικέ πολιτικέ οι τεχνικές παραγωγής καλύπτουν ένα φάσμα ευρύτερο σε σχέση με την απλή παραγωγικότητα, δεν θα θέσει αυτό σε κίνδυνο την κοινή γεωργική πολιτική. Η απώλεια των μέσων που στηρίζουν την κοινή γεωργική πολιτική μπορεί να πλήξει την βιωσιμότητα καθώς και την ανταγωνιστικότητα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα ήθελα να κάνουμε μια επισκόπηση, σύντομη επισκόπηση ε, σχετικά με την ανακοίνωση. Τι περιμένει η κοινωνία από τη γεωργία, η υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα, καλύτερη χρήση των ε, φυσικών πόρων, ε, σωστότερη χρήση των καλλιεργούμενων γεών, χωρίς να παραβλέπουμε τις ανάγκες κανενός. Αυτές οι προσδοκίες δεν είναι νέες, προβλέπονται εξάλλου και στη συνθήκη ε, ακόμη και στη νέα συνθήκη της ε, Λισαβόνας για την ανταγωνιστικότητα η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με την μεταρρύθμιση του 1992 μόνο που σήμερα η ανταγωνιστικότητα σημαίνει πολλά περισσότερα ε, από την παραγωγικότητα. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να διευρύνουμε λίγο την έννοια και αυτό είναι ο στόχος της μεταρρύθμισης που εισηγούμαστε σήμερα. Ε, πρέπει να υπενθυμίσουμε επίσης ε, ότι προετοιμάζουμε αυτή την μεταρρύθμιση στα πλαίσια της διευρυμένης Ευρώπης. Πρώτη φορά προβαίνουμε σε μεταρρύθμιση μετά τη μεγάλη διεύρυνση της Ένωσης προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Πρώτη φορά 27 κράτη-μέλη συζητούν αυτή τη μεταρρύθμιση και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, διότι όπως σας είπα έχουμε ενώπιόν μας ένα νέο τύπο γεωργίας ε, δεδομένης της διεύρυνσης. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι επίσης ένα σημαντικό, μια σημαντική συνιστόσα, όπως σας έλεγα προηγουμένως, της ε, στρατηγικής Ευρώπης 2020 και βασικό μέσο για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της στρατηγικής. Με ποιο τρόπο λοιπόν ε, προτείνουμε να επιτευχθούν αυτοί οι προαναφερθέντες στόχοι. Πρώτα απ' όλα, ε, με την ε, νέα δομή δύο πυλώνων ε, οι ενισχύσεις του εισοδήματος παραμένουν αναγκαίες αλλά πρέπει να είναι πιο στοχευμένες και πιο δίκαιες. Αυτό συμπεριλαμβάνουμε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Επίσης να καλύψουμε τις ανάγκες των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που πρέπει ε, να συμβάλλουν στον όλο διάλογο για την ε, χωροταξική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι εκμεταλλεύσεις αυτές ανταποκρίνονται, μάλλον απευθύνουν σε διάφορες αγορές, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί έχουν σημειωθεί οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμη. Επίσης, πρέπει να στηρίξουμε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο, δηλαδή τους ενεργούς γεωργούς, πρέπει να ορίσουμε αυτή την έννοια Επίσης, για να είμαστε πιο ρεαλιστές ε, και πιο αξιόπιστοι με τις άμεσες ενισχύσεις, ε, προτείνουμε ε, θέση ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις. Επί τη βάση της εξής αρχής θα πρέπει να στηρίζετε το εισόδημα αυτών των γεωργών. Δηλαδή, από ένα επίπεδο ενίσχυσης και μετά δυσκολευόμαστε να αιτιολογήσουμε μια ενίσχυση ως ενίσχυση του εισοδήματος. Γι' αυτό και θέτουμε το ανώτατο όριο και αυτό συνδέεται με το ρόλο ε, των μικρών αλλά και των μεγάλων εκμεταλλεύσεων, γιατί οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις στηρίζουν την απασχόληση. Λοιπόν, ε, αυτές οι επενδύσεις του πρώτου πυλώνα ε, προτείνουμε τις άμεσες ενισχύσεις να τις χρησιμοποιήσουμε μέσω κινήτρων, παραδείγματο χάρη, που θα εξασφαλίσουν τη διαχείριση των φυσικών πόρων, να μην συνιστούν μόνο δεσμευτικό στοιχείο πλέον. Ποιε είναι οι προτάσει για να καταλάβετε ποιο προσανατολισμό ε, προτείνουμε, ποια είναι αυτά τα κίνητρα, ποια είναι τα μέτρα που προτείνουμε για να έχουμε μια ε, πρόσθετη στήριξη γεωργή. Δεν πρόκειται για μέτρα που οδηγούν σε αύξηση του κόστους ε, για τον παραγωγό. Άμυψη σπορά, παραδείγματο χάρη διατήρηση μονίμων βοσκοτοπιών, αγρανάπαυση, άλλα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Δεν οδηγούν αυτά σε αύξηση του κόστους αυτό αυτόματα, αντίθετα οδηγούν σε πιο βιώσιμη, πιο ανταγωνιστική ε, γεωργία. οι λιγότερο ευνοούμενες περιοχές. Τι γίνεται, στον πρώτο πυλώνα προτείνουμε τα κράτη-μέλη να μπορούν να έχουν μια ενισχυμένη στήριξη πέρα από τη βασική ενίσχυση, δηλαδή για τους γεωργούς των λιγότερο ευνοούμενων περιοχών, κρατώντας όμως τις ειδικέ ενισχύσεις με εθνική ε, συγχρηματοδότηση. Αυτό στο δεύτερο πυλώνα. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Ε, ας περάσω στο δεύτερο πυλώνα. Ο στόχος είναι να προσφέρουμε εργαλεία μέσα ε, που θα κατοχυρώσουν αυξημένη ανταγωνιστικότητα, ε, ε, καλύτερη διαχείριση φυσικών πόρων και εδαφών, με μέσα όμω που προσφέρουν ευελιξία, που προσφέρουν ένα περιθώριο ελιγμών στα κράτη-μέλη, ε, γιατί θα κάνουν επενδύσει από το δικό του προπολογισμό για την κατάρτιση. Δηλαδή, θα στοχευμένα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ή στοχευμένα μέτρα για τι λιγότερο ευνομένε περιοχέ και μέτρα που προωθούν την τοπική, τις τοπικές πρωτοβουλίες περί καινοτομίας. Το θέμα των, ε, της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών θα είναι ένα γενικό θέμα του δευτέρου πυλώνα με δείκτες που θα προτείνουμε ούτως ώστε οι δράσεις που θα στηριχθούν ε, βάσει του δεύτερου πυλώνα να έχουν και αυτή τη διάσταση, δηλαδή να καταπολεμούν και τις ε, κλιματικές αλλαγές. Ε, σας διαβεβαιώ ότι όταν σας μιλάω για τις τοπικές πρωτοβουλίες καινοτομία, θέλουμε να βασιστούμε στην εμπειρία των προγραμμάτων LEADER και να διευρύνουμε την εμπειρία αυτή και σε άλλες πρακτικές που αφορούν ειδικότερα ίσως τον γεωργικό τομέα. Προτείνουμε επίσης στο δεύτερο πυλώνα να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τους διάφορους τρόπους ε, θέσης εμπορία ε, που θα προσαρμόζονται ε, σε διάφορα είδη γεωργίας, δηλαδή βραχία κυκλώματα, παραδείγματος χάρη τοπικές αγορές, γιατί για την τροφική αλυσίδα μπορούμε να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τα μεγάλα συστήματα διανομής που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ε, για τη διαχείριση τώρα των μέσων της αγοράς, ε, ούτως ώστε να στηρίξουμε τα εισοδήματα των γεωργών. Αυτό είναι θέμα του δευτέρου πυλώνα και χρησιμοποιούμε την ιδιαιτερότητα του πρώτου και του δευτέρου πυλώνα. Δηλαδή, ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε δίχτυα ασφαλείας με κάποια από αυτά τα μέσα θέλουμε να δρούμε ε, ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά, να ενεργοποιούμε ε, ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά αυτά τα μέσα και πέραν αυτού προτείνουμε το δεύτερο πυλώνα για να έχουμε αυτή την πολιετή και πιο ευέλικτη προσέγγιση. Μέσα δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε την ε, μεταβλητότητα των εισοδημάτων μέσα από ε, ασφαλιστικά συστήματα, ταμεία αμοιβαίας βοήθειας, ε, όπως αυτά τα αισθήματα που ήδη ισχύουν σε κάποια κράτη-μέλη για τους γεωργούς. Για τη διαχείριση των αγορών και την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας των εισοδημάτων είναι θέματα επιτάπητος που δεν καλύπτονται άμεσα από αυτό το σχέδιο μεταρρύθμισης. Ε, διότι υπερβαίνουν το ειδικό θέμα της γεωργίας. Είναι ζητήματα που θα πρέπει να ενταχθούν σε γενικότερη ανάλυση της ε, ε, αγροπεριβαλλοντικής αλυσίδας με τον, με τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη τον Επίτροπο Νταλή συζητήσαμε πριν από λίγες μέρες ε, τις αλλαγές ε, που θα προκύψουν στις προσεχείς ε, μήνες και επίσης θα, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις σε διεθνέ επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι η Γαλλία θα αναλάβει την προεδρία της ομάδας G20 και θα επιληφθεί αυτού του ζητήματος και θέλουμε φυσικά να συμβάλλουμε στο διάλογο. Αυτή είναι η πολιτική θεώρησή μας για την κοινή γεωργική πολιτική του μέλλοντος. Η πολιτική αυτή πρέπει να επιτρέπει γεωργούς να να, να ιδρύουν επιχειρήσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τη αγοράς και της ε, κοινωνίας. Η γεωργία θέλουμε να είναι πυλώνα στήριξη ε, της υπαίθρου. Α μην είμαστε αφελεί. δεν γίνεται αυτό χωρίς ε, την χρηματοδοτική στήριξη του κράτους, του δημοσίου τομέα. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε επαρκή ε, εθνική ε, ε, χρηματοδοτική στήριξη και ελπίζω ότι εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας αλλά και μέσω των δραστηριοτήτων που έχετε στις διάφορες πολιτικές ομάδες και σε άλλες συναρμόδιες επιτροπές θα συμβάλλετε στην ε, κατάρτιση ενός ε, συνεκτικού ε, μεταρρυθμιστικού σχεδίου που θα ακολουθεί αυτούς τους ανατολισμούς που σα εξέθεσα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερος κύριε Επίτροπε και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων στον καθένα για τρία λεπτά. Εν συνεχεία θα έχουμε τις απαντήσεις του Επιτρόπου και θα περάσουμε μετά στη συζήτηση όπου θα μπορεί να λάβει το λόγο οποιοδήποτε άλλο μέλος Επιτροπής μας εφόσον το επιθυμεί έχοντας στη διάθεσή του δύο λεπτά. Σας παρακαλώ όλοι να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευσης για να μπορέσει ο Επιτρόπος να απαντήσει. Λοιπόν, αρχίζει η συζήτηση και θα δώσω τώρα το λόγο στο συντονιστή της ομάδας του και επόμενος Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ανακοίνωση αυτή που μας έκανε και τη μία ημέρα καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, θα την αντέξουμε. Οι ανακοινώσει για την κοινή γεωργική πολιτική για το 2013 αποτελεί μια σημαντική βάση των συζητήσεων για τις ε, εργασίες που θα ακολουθήσουν στο Κοινοβούλιο τις επόμενες ε, μήνες. Κοιτάμε την μεταξέλιξη της κοινή αγροτικής πολιτικής μετά το 2013 και θεωρώ ότι με την ανακοίνωση αυτή ως Κοινοβούλιο μπορούμε να αξιοποιήσουμε πολλές δυνατότητες που έχουμε για τις ε, προτάσεις που μας γίνονται προκειμένου να τις συμπεριλάβουμε και να τις αναπτύξουμε με λεπτομέρεια στις εκθέσεις μας. Πολλά αναφέρεται λοιπόν κατά αποκοπήν στην ανακοίνωση. Το δύσκολο θα είναι αυτά τα στοιχεία να μετατραπούν σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Γιατί ξέρετε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και πολλά θα χρειαστεί να συζητήσουμε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτή των προτάσεων. Καλώς ορίζω ιδιαίτερα κύριε Επίτροπε το γεγονός ότι κρατάτε στην πρότασή σας το μοντέλο αυτό των δύο πυλώνων και θα ήθελα να σας πω θα πρέπει να διαμορφωθεί και στην πραγματικότητα. Θα πρέπει φυσικά να περιοριστούν και τα διοικητικά, το διοικητικό βάρος. Αλλά την πρώτη φορά που διάβαζα ε, εκ πρώτης όψεως η ανακοίνωση με κάνει να πιστεύω ότι δεν θα καταλήξουμε σε πιο περιορισμένο διοικητικό άχθος, αλλά σε πιο έντονο. Και η εντύπωση που μου δίδεται είναι ότι τα μέτρα θα πρέπει να εκφραστούν λεπτομερώς σε ό,τι αφορά τον πρώτο πυλώνα για να περιοριστεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση. Γενικά συμφωνούμε ότι είναι καθήκον της ε, Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής να εξασφαλίσει την επιστηστική ασφάλεια και για το μέλλον σε ό,τι αφορά το μισό δισεκατομμύριο πολίτες που έχουμε. Και στο σημείο αυτό Είμαι αισιόδοξο ότι το Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει το ρόλο του. Είμαι αισιόδοξο και σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει με τι άλλε ομάδε. Θα καταθέσουμε προσπα... Ε, προτάσει για το πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την μελλοντική επιστημιστική ασφάλεια. Θέλουμε να προτείνουμε και κάποιε προσθήκε. Το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο πριν από κάποιο καιρό αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία σε ό,τι αφορά το διεθνές εμπόριο και τις εισαγωγές από τρίτα κράτη-μέλη θα πρέπει να τηρούνται τα δικά μας πρότυπα ποιότητας σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή, των ζώων. Θα προσθέσουμε λοιπόν σημαντικά στοιχεία ως κοινοβούλη, τα οποία θα συμπληρώσουν την ανακοίνωση αυτή. Γιατί αν υπάρξουν νέες προτάσεις με το Συμβούλιο, με, το, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα διαπραγματευτούμε προκειμένου η αγροτική πολιτική, το ευρωπαϊκό μοντέλο που θέλουμε να αναπτύξουμε, να μην καταστεί υπερβολικά σχολαστικό και υπερβολικά γραφειοκρατικό. Και νομίζω ότι πολλά θα έχουμε να κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εισηγητής για το θέμα αυτό και είμαι βέβαιος ότι με θετικό τρόπο θα επεξεργαστούμε την ανακοίνωσή σας εδώ στο Κοινοβούλιο προκειμένου να καταλήξουμε σε μια σωστή πρόταση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τες. Α, μετά τον κύριο Τες, ο κύριος Σάντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσίαση της πρότασής του. Ε, έχουμε ελπίδες ε, και είμαστε με μετριοπαθώς αισιόδοξοι σε σχέση με τη μεταρρύθμιση. Μα παρουσιάσατε το όραμά σα και διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι πολλέ από τι ε, προτάσει που έκανε τον Απρίλιο ε, οι σοσιαλιστέ ε, συνάδουν με την ανακοίνωση τη επιτροπή. Συμφωνούμε με αυτά που είπατε για τι προκλήσει και του στόχου, διατροφή, επιστημιστική ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντο, παραγωγή βιώσιμων τροφίμων, βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, ισόρροπη ανάπτυξη

όλων των περιφερειών ε, ε, και πραγματικά σε σχέση ε, με τα, ιστορικά κριτήρια και τα κριτήρια κατανομής των ενισχύσεων, τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, την ανησυχία που είπατε να έχουμε δηλαδή μεγαλύτερη δικαιοσύνη για την κατανομή της συγχρηματοδότησης ανάμεσα στην Ένωση και τα κράτη-μέλη, τα κίνητρα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τα νέα μέσα για τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων, το ανώτατο όριο για τις ε, ενισχύσεις ε, και όλα αυτά τα μέτρα στα οποία δεν θα επισέλθω ε, θα σα προσφέρουμε τη στήριξή μας. Έχουμε βέβαια και κάποιες δυσκολίες με άλλα στοιχεία που αναφέρατε. Λυπούμε θα παραδείγματος χάρη που ο τομέας της απασχόλησης δεν αναφέρεται ρητά ως κριτήριο για τη χορήγηση των ενισχύσεων. Θεωρούμε ότι η πρόταση, ε, δεν υπάρχει αντιστοιχεία για αυτό που εξαγγείλατε ότι θα επικρατήσει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και τα μέτρα που προτείνατε για να επιτύχουμε αυτό τον στόχο ε, θεωρούμε επίσης ότι δεν λάβατε επαρκώς υπόψη ε, το θέμα τη του ε, των ενισχύσεων στο γαλακτοκομικό τομέα μέχρι το 2015. Θα πρέπει να σταθμίσετε αυτό το θέμα της πάυσης των ενισχύσεων. Δεν πρέπει να θεωρείτε δεδομένο ότι θα διακοπούν οι ενισχύσεις το 2015. Έχουμε ενδιασμούς και θα θέλαμε να διευκρινίσετε και κάποια άλλα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, αυτή αυτή η έννοια του ενεργού γεωργού. Ε, ε, είναι στο άρθρο 28 ε, του κανονισμού 73-2009 για το health check. Ε, τι μας προτείνετε, να είναι υποχρεωτική αυτή η έννοια και να μην επαφίεται στην διακριτικότητα, στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Επίσης μιλήσατε για απλουστευμένο σύστημα ενίσχυσης των μικρών εκμεταλλεύσεων. Πώς θα ορίσουμε τον μικρό γεωργό, εσείς θέλετε να εισαγαγείτε αυτή την έννοια χωρίς να το διευκρινίζετε και είπατε θα το χρησιμοποιήσετε για την σταθεροποίηση των εισοδημάτων. Τέλο, μέσα στο κείμενο υπάρχει ένα στοιχείο που μα δημιουργεί σοβαρού ενδιασμού ε, και διάβασα πολλέ φορέ αυτή τη φράση και δεν την κατάλαβα. Πρέπει, λέτε, να θεσπίσουμε ένα σύστημα που ε, περιορίζει τα κέρδη και τι απώλειε των κρατών μελών, εγγυούμενοι ότι σε όλου του τομεί οι γεωργοί, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα λάβουν ένα κομμάτι από ε, το ελάχιστο εγγυημένο συγκεκριμένο μέσο εισόδημα. Ε, ε, δηλαδή αυτοί που παίρνουν περισσότερο θα παίρνουν λιγότερα, αυτοί που παίρνουν λιγότερο, λιγότερα μπορούν να λάβουν υψηλότερες ενισχύσεις. Οι γεωργοί θα λαμβάνουν ε, ένα κομμάτι, ένα τμήμα, ένα ελάχιστο τμήμα του μέσου, ε, της μέσης ελάχιστης ενίσχυσης. Μα τι εννοείται, είναι κεντρικό στοιχείο της παρούσας μεταρρύθμισης και αυτή η διατύπωση είναι εξαιρετικά συγκεκριμένη. Σας παρακαλούμε λοιπόν ε, διευκρινίστε το περιεχόμενο αυτής της ε, πρότασης. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λουίς George Λάιεν από την ομάδα των Φιλελευθέρων. Thank you, uh, President. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα συμφωνήσω με τα σχόλια των συναδέλφων συντονιστών σας καλωσορίζω και εγώ στην Επιτροπή μας. Χαιρετίζω και την ανακοίνωση που μας εκθέσατε αναφέροντας ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον και την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γεωργίας κατά τα προσεχή έτη. Το έγγραφο σαφώς ε, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα και όλοι κάτι θα βρουν για να ε, καθησυχαστούν ότι τουλάχιστον έχετε ακούσει προσεκτικά εσείς τι έχει υποθεί μέχρι τώρα στη συζήτηση. Τώρα, η μεγάλη ευκαιρία που έχουμε εμεί στην Επιτροπή μα που θα πρέπει να επεξεργαστούμε αυτό το νομοθέτημα ουσιαστικά είναι να δώσουμε μια εστίαση και μια μεγαλύτερη σαφήνεια στα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για του Ευρωπαίου αγρότε και βέβαια για να φέρουμε σε πέρα και το δικό σα όραμα για ένα βιώσιμο και ευημερούν σύστημα γεωργία και στο μέλλον. Σίγουρα στόχο είναι η παραγωγή πρώτη ποιότητα ε, τροφίμων που θα καταλήγουν στο πιάτο μα, στο πιάτο των Ευρωπαίων καταναλωτών. Χαιρετίζω αυτό που είπατε για την δίκαιη αμοιβή επίσης για το ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των τροφίμων. Να γνωρίζω επίσης ότι τα κίνητρα που λέτε ότι πρέπει να υπάρχουν ανταμοιβέ και βέβαια και η, βιωσιμότητα που θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης αυτής. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ε, το οποίο αναφέρατε και εσείς και τονίσατε. Σε ό,τι αφορά το τέλος ε, των ιστορικών ε, πυρωμών, μάλλον είναι η σωστή κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να ε, βαδίσουμε και η συμπερίληψη των μειονεκτικών περιοχών στον πυλώνα 1. Έχω κάποια ερωτήματα πάνω σε αυτό, κάποια ερωτηματικά μάλλον. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε τα εξής. Χαιρετίζομαι τη συμπερίληψη των μειονεκτικών περιοχών ως ε, προτεραιότητα στις πληρωμές του πυλώνα 1. Πώς θα λειτουργήσει ακριβώς αυτό όμως. Θα έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να έχουν ξεχωριστό πρόγραμμα για τις, λιγότερο ευνοούμενες ε, ευνοϊκές περιοχές στο πλαίσιο των πληρωμών και είπατε ότι θα περάσουμε από το ιστορικό ε, σύστημα αυτό του υπολογισμού και καταβολής των πληρωμών σε ένα άλλο σύστημα. Πότε θα γίνει αυτό, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας, γιατί είναι προφανές ότι είναι ένα ιδιαίτερα δυσχερές ζήτημα και θα δημιουργήσει και προβλήματα σε πολλά κράτη-μέλη. Μιλήσατε επίση για το πρασίνισμα των άμεσων πληρωμών. Εγώ το χαιρετίζω αυτό. Παρ' όλα αυτά έχω κάποιε ανησυχίε. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην έκθεση την οποία συνέταξα μάλιστα εκ μέρους ε, της Επιτροπής και στις συζητήσεις που είχαμε ήταν σαφές ότι αν δεν προσέξουμε θα καταστήσουμε μη ανταγωνιστική την Ευρωπαϊκή Γεωργία και αυτό πρέπει να είναι σαφές. Το πρασίνισμα των άμεσων πληρωμών πρέπει να αφορά την βιωσιμότητα, την αύξηση της αποδοτικότητας και όχι στην μείωση της ανταγωνιστικότητας. Και ένα άλλο ερώτημα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της νομοθετικής πρότασης τι κάνετε με τις αποφάσεις περί, δημοσίων, περί προϋπολογισμού. Γιατί σίγουρα το ένα επηρεάζει το άλλο. Και πώς μπορεί κανείς να προχωρήσει σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις αν δεν γνωρίζει ακριβώς ε, το προϋπολογισμό που θα έχει στη θέση του. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ τον ε, George Lyon, ο James Ingleson. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ να συμφωνήσω με του υπόλοιπου οι οποίοι καλωσόρισαν ε, το έγγραφο, την ανακοίνωσή σα επιτέλου τη λάβαμε, γιατί αναφέρει πολλά στοιχεία. Και επιτέλους ε, ακούμε τι σκοπεύετε να κάνετε μακροπρόθεσμα. Όλοι ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε πρώιμη φάση της διαδικασίας αυτής, η οποία θα συνεχιστεί, φαντάζομαι, και θα καλύψει και τα επόμενα δύο έτη σε κάποιο βαθμό είναι καλό το έγγραφο αυτό γιατί μας αναφέρει αυτά που ήδη ξέρουμε. Και τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα μεταξελιχθεί το έγγραφο αυτό προκειμένου να διαμορφωθεί με τρόπο εφαρμόσιμο επιτόπου για τον κάθε αγρότη. Αν θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω ποιες είναι οι θέσεις σας σε ό,τι αφορά την έννοια του ενεργού γεωργού γιατί πολύ καιρό ακούμε την έννοια αυτή, τον ορισμό αυτό. Αλλά ποιος είναι τελικά ο ενεργός ε, γεωργός. Είναι ο γεωργός ο οποίος δουλεύει επί τόπου. Ο δικηγόρος δηλαδή που πάει και αγοράζει ένα μικρό αγροτεμάχιο είναι ενεργός γεωργός. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η συζήτηση και θα πρέπει να την κάνουμε. Επίσης μιλάτε για την προσπάθεια συγκράτηση των τιμών. Έχετε ε, κάποια ιδέα ποιο θα είναι το ανώτατο όριο, ποιο θα είναι το πλαφόν. Γιατί νομίζω ότι από πολλές απόψεις θα είμαστε κατά ίσως ε, της ρύθμισης αυτής. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την πολλαπλή συμμόρφωση, για παράδειγμα. Πρέπει να πω, Επίτροπε, και διαβάζω και ακούω πολλές φορές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες που ακολουθούμε. Κι όμως κάθε φορά που κάτι προσπαθούμε να απλοποιήσουμε τελικά δημιουργούμε πιο πολύ γραφειοκρατία και άλλες επιθεωρήσεις και άλλους ελέγχου και άλλους προορισμού για του αγρότε. Επίση, να μα πείτε δύο λόγια παραπάνω, γιατί κάτι πολύ σημαντικό που μου το θέτουν και πάρα πολλοί γεωργοί είναι ότι πάρα πολλοί γεωργοί λαμβάνουν πάρα πολλές μικρές βοήθειες από τα ταμεία. Πώς ορίζεται λοιπόν ο μικρός γεωργός. Και θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο σε ό,τι αφορά αυτό το πρασίνισμα. Πολλές ε, τροπολογίες θα κατατεθούν τα επόμενα, τους επόμενους μήνες, είμαι βέβαιος. Πρόεδρε, να κλείσω λέγοντας το εξή. Θεωρώ αδιάσυστα ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να είναι γεωργική πολιτική, πολιτική για τη γεωργία, για την ασφάλεια του εφοδιασμού των τροφίμων δεν είναι κοινωνική πολιτική ούτε περιβαλλοντική πολιτική, αλλά να είμαι σαφή ότι πιστεύω ότι παρά το γεγονό ότι δεν είναι περιβαλλοντική πολιτική, η γεωργική πολιτική και οι γεωργοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλλουν με σημαντικό τρόπο για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο, για την προστασία του περιβάλλοντο και το κάνουν ήδη. Αλλά μπορούν να κάνουν και παραπάνω αν έχουν την ευκαιρία. Αλλά να μην μείνουν αμέτωχοι, γιατί αυτή είναι τελικά που θα πρέπει να εξασφαλίσουν την εμπιστευτική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο Τζέιμ. Ο Μάρτιν Χόσλιν, Πρόεδρε, Επίτροπε. Επίτροπε να σα ευχαριστήσω καταρχάς για το γεγονό ότι έρχεστε πρώτα-πρώτα στο Κοινοβούλιο για να παρουσιάσετε την πρότασή σα και όχι σε άλλου. Είναι μεγάλη χειρονομία και την εκτιμούμε. Μας θέσατε τα σωστά ερωτήματα και κάνατε πολλές αναφορές για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί στο μέλλον η ΚΑΠ. Να σας πω ότι σας υποστηρίζουμε σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμιστικές σας προτάσεις, γιατί νομίζω πολλά στοιχεία αναφέρετε τα οποία μας βρίσκουν σύμφωνους. Με απότερο σκοπό να πρασινίσει η αγροτική πολιτική συσσαγωγικά αλλά να διαμορφωθεί και στο διεθνές προσκήνιο γιατί όλους αυτούς τους στόχους θα πρέπει να τους έχουμε υπόψη στην αγροτική μεταρρύθμιση προκειμένου να γίνει αποδεκτή και από την κοινωνία. Δεν είναι μόνο για τους γεωργούς η μεταρρύθμιση αυτή, αλλά είναι και κοινωνικό θέμα. Θα πρέπει να υπάρχει και μια κοινωνική βάση. Θα πρέπει ο φορολογούμενος να θεωρεί ότι υπάρχει απόδοση της επένδυσης αυτής, για παράδειγμα. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια ανταπόδοση. Και σωστά είπατε, τύφονται θέματα όπως η προστασία, η βιοπικιλότητα, ποιε είναι οι απαιτήσει της κοινωνίας, στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί επιτέλους η γεωργία. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν τη σωστή τεκμηρίωση, τη σωστή βάση, τη σωστή δικαιολόγηση των χρημάτων που δαπανούνται. Και στο θέμα της δικαιοσύνης ε, θέτεται πολύ σημαντικά και σωστά ε, ζητήματα και σε ό,τι αφορά το, τη συγκράτηση των τιμών. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Υπάρχει ένα θέμα αδικαιοσύνης μεταξύ των κρατών ε, μέλων, αλλά φυσικά αυτό αφορά κυρίως το εσωτερικό της, ε, του γεωργικού κλάδου. Σε, θα πρέπει να εστιαστούμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα αυτά τα ε, λέμε, αλλά υπάρχει πραγματικά μια ανισότητα σε ό,τι αφορά τις πληρωμές και αυτό θα πρέπει επιτέλους να το διορθώσουμε. Τι είναι το βασικό πρίμα επίσης. Και επίσης θα πρέπει να εστιαστούμε στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Όλα αυτά τα αναφέρεται στην ανακοίνωση και οι θέσει εργασίας αποτελούν ένα βασικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τη μελλοντική να δούμε και τι συμβαίνει με τις πληρωμές, αλλά βλέπουμε και την συνολική ε, οπτική. Και να διευκρινίσω το εξής, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να δούμε ε, να μην στρεβλώνουμε το διεθνές εμπόριο. 80 έως 85% των αναγκών μας καλύπτονται με εισαγωγές. Και φυσικά είμαστε κι εμεί συνυπεύθυνοι αν εξαφανίζονται τα τροπικά δάση στη Βραζιλία. Αλλά κάτι επίση πολύ σημαντικό είναι, είναι το ισοζύγιο μεταξύ της γεωργία και του εμπορίου. Το θίξατε το θέμα αυτό και είναι σαφέ ότι θέλουμε να ισοσκελιστούν τα δύο αυτά στοιχεία. Θα πρέπει να πάρουν μεγαλύτερο τμήμα. Γεωργή, Τώρα, το θέμα του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα είναι πολύ ενδιαφέρον και θα πρέπει να δούμε πώς θα δημορφωθεί η ισορροπία. Είπατε ότι υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις και στην τελική ανάλυση θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η κατανομή μεταξύ των δύο πυλώνων για να υπάρχει περιθώριο και για την αγροτική ανάπτυξη. Αυτά τα ερωτήματα μένουν ανοιχτά. Και τώρα το μπαλάκι έχει έλθει στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει με θάρρος και με θέληση να προβούμε σε μεταρρυθμίσεις, να καταπιαστούμε με τα θέματα αυτά και είμαι βέβαιος ότι θα καταστεί αποδεκτή η πρότασή σας. Ευχαριστώ Μάρτιν, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει ο Λορέντσο Παντάνα. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και εγώ με αυτούς οι οποίοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στον Επιτρόπο για την παρουσίαση του εγγράφου αυτού. Πολλά σημεία του τα συμμεριζόμαστε. Είναι το αρχικό βέβαια έγγραφο, στη συνέχεια θα δούμε. Θα δούμε τα πιο συγκεκριμένα σημεία, τις πιο συγκεκριμένες πτυχές. Πάντως ένα πάρα πολύ ε, σαφές ε, είναι, είναι, είναι το εξή, ότι υπήρξαν προβλήματα κατά το παρελθόν γιατί η κοινή γεωργική πολιτική έχασε ένα μέρο τη αξιοπιστία τη. Αν δεν υπάρχει όμω κοινή γεωργική πολιτική, απειλείται η ίδια η επιβίωση της γεωργίας όπως τη γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι ορισμένοι να μην έχουν την βούληση για να δώσουν τα απαραίτητα κονδύλια για τη γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν περισσότερα πράγματα, διότι αν δεν υπάρχει ο επαρκή προπολογισμό, είναι προφανέ ότι όλε οι άλλες ε, πολιτικέ, όπω είπε και ο Τζίμι Νίκολσον, δεν θα μπορούν να έρθουν σε πέρα. Ε, Παραδείγματο χάρη και για την κτηνοτροφία χρειάζεται μια πολιτική. Και σίγουρα καλά και άγια όσα κάνουν οι αγρότες ε, και οι κτηνοτρόφοι για τη βιωσιμότητα. Πώ όμω θα του επιτρέψουμε να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους αυτές. Και πραγματικά νομίζω ότι διακυβεύονται πολλά για τους ίδιους τους αγρότες ε, ε, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Δηλαδή και οι ίδιοι ε, θέλουν την προστασία του περιβάλλοντος. Και σίγουρα πρέπει να συνεργαστούμε με τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό που δεν θέλουμε ε, δεν είναι να τους δίνουμε χρήματα μόνο, αλλά να τους βοηθήσουμε να διατηρήσουν ε, την ανταγωνιστικότητά τους και την απασχολησιμότητά τους. Διότι υπάρχει κόσμος ο οποίος απασχολείται στην ε, γεωργία. Είναι ένα αρκετά σημαντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού το θέμα της ε, διακύμανσης ε, του εισοδήματος αυτό δεν νομίζω ότι το βλέπουμε όπως θα έπρεπε στην ανακοίνωση. Και πρέπει να δούμε και το ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο τη γεωργία. Δηλαδή σε ορισμένες χώρες ε, υπάρχουν εισαγωγές γεωργικών προϊόντων τα οποία δεν πληρούν, σε ό,τι αφορά την παραγωγή τους, τα κριτήρια που πληρούν οι δικοί μας αγρότες εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα αυτό ενθαρρύνει και τη διακύμαση των τιμών, και δημιουργεί και άλλα ζητήματα. Αν λοιπόν δεν ε, αναλάβουμε δράση θα έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Είπατε επίσης ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις τοπικές πρωτοβουλίες και αυτό είναι πολύ θετικό για μένα γιατί είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της γεωργίας. Η γεωργία μπορεί να χρησιμοποιεί το τοπικό εργατικό δυναμικό, τα τοπικά προϊόντα και αυτό είναι μια, ένα από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Καλό είναι που συζητούμε για τη γεωργία. Ε, σίγουρα έχει χάσει μέρος αξιοπιστίας στη συγκεκριμένη πολιτική. Μπορούμε όμως κάπως να την αποκαταστήσουμε κύριος Λε Γιάρικ. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε. Ευχαριστούμε για τις εργασίες διαβούλευσης που προηγήθηκαν ε, της δημοσίευσης και παρουσίας της ανακοίνωσης. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία επαναπροσανατολισμού της πολιτικής μέσα στο εγγραφό σας, ε, επαναπροσανατολισμού δηλαδή της γενικότερης φιλοσοφίας που διέπει την κοινή γεωργική πολιτική. Αυτή η έννοια του ενεργού γεωργού νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την κατανομή των ενισχύσεων. Το θέμα, η πρόκληση του το ανωτά του ορίου επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ενισχύσεις. Τα κίνητρα τα μέτρα κίνητρα για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν επίσης σημασία. Όλα αυτά που μας είπατε για την ευελιξία, όλα αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα και δεν ξέρω αν έχετε κάποιες πρώτες απαντήσεις να μας δώσετε. Όπως ε, προείπαν και οι συνάδελφοι, ε, αναρωτιόμαστε, ε, είμαστε σίγουροι ότι θα διατηρηθούν τα κονδύλια όσοι έχουν μέσα στον προϋπολογισμό. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σχετικά με αυτό. Επίσης, δεν αναφερθήκατε καθόλου και καταλαβαίνω γιατί, διότι το έχουμε συζητήσει το θέμα στο παρελθόν, δεν μιλήσατε για τους μηχανισμούς προστασίας της γεωργίας μας. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός προστασίας, και είπατε και αντιλαμβάνομαι ε, τι εννοείτε, ε, ε, για την βιωσιμότητα και την, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ε, καταλαβαίνω αυτό που είπατε αν δεν έχουμε συστήματα προστασίας σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία, όπως έχει σήμερα δηλαδή, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Οι ε, εργασιακοί κανόνε, οι περιβαλλοντικοί κανόνες διαφέρουν από μια χώρα σε άλλη και τελικά πλήττεται η γεωργία λόγω της ανταγωνιστικότητας. Και δεν σας μιλάω για την ανταγωνιστικότητα στο ιστορικό τη Ένωση, ε, διότι δεν πιστεύω δεν πιστεύω ότι υπάρχει μία μόνο ευρωπαϊκή γεωργία. Είναι διαφοροποιημένη, έχει πολλαπλές διαστάσει και αυτό πρέπει να ισχύει ούτω ή άλλω. Τώρα, αυτά που μας προτείνεται τελούν υπό δύο αιρέσει. Πρώτον, ε, ε, ο, το, το τέλος του κύκλου διαπραγματεύσεων της Ντόχα. Ε, έχετε στοιχεία γι' αυτό. Επίσης, διμερείς συμφωνίες. Όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, εάν συνάψουμε αυτή τη συμφωνία με τη Μερκοσούρ για την εισαγωγή βοήου κρέατος, αυτό συνεπάγεται καταστροφή για ολόκληρες περιοχές της Ένωσης, ε, κυρίως στο Μασίφ Σαντράλ ε, στη Γαλλία. Γνωρίζετε πολύ καλά αυτή την περιοχή. θα πρέπει να προβλέψετε ένα μηχανισμό προστασίας που θα είναι επωφελής για όλους, ε, διότι ε, μιλάμε για το περιβάλλον. Αναφερθήκατε πολλαπλώς στο περιβάλλον και ορθώς. Στην παραγωγή των πρωτεϊνών ε, της σόγιας, παραδείγματος χάρη, τι κάνουμε, εξάγουμε την μόλυνση σε άλλες χώρες για να έχουμε παραγωγή χαμηλού κόστου και για να δεν έχουμε επάρκεια στις πρωτενε. Κάτι άλλο τώρα. Αντιλαμβάνομαι ε, ποιο είναι ο στόχο σα με το δίχτυ ασφαλεία, με το ελάχιστο επίπεδο παρέμβαση, τούτου λεχθέντο δεν ε, είμαστε αρκετά φιλόδοξοι, κυρίως ε, για την ελάχιστη τιμή. Αν αυτή την ελάχιστη τιμή τη συνδέσετε με το ανώτατο όριο των ενισχύσεων, ε, θα έχετε μια πολύ καλή ιδέα, διότι ταυτόχρονα έχουμε και απελευθέρωση, κυρίως όταν μιλάμε για την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Καταλαβαίνετε ότι η γεωργία μας θα αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνισμό και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ε, επίτροπε, ακούσατε όλου τους συντονιστέ από όλε τι πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για μια πρώτη αντίδραση και μετά θα προβούμε στη συζήτηση. Ο Επίτροπος έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι στο δυνατόν ε, πιο γρήγορος, αλλά ταυτόχρονα βέβαια να σας δώσω και κάποια διευκρινιστικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, ιδιαίτερος γενική προσέγγιση το περίμενα. Περίμενα να ακούσω ότι αν ένα έγγραφο είναι συνεκτικό, ε, ουσιαστικά ε, πρόκειται για μια πολύ γενική προσέγγιση. Αν είχα έρθει με πολλέ λεπτομέρειε, θα μου λέγατε, μα δεν μα αφήνετε τα περιθώρια, κύριε Επίτροπε, να διατυπώσουμε τι προτάσει μα. Πρότεινα λοιπόν κάτι γενικό, διότι ο ρόλο του εγγράφου είναι ακριβώ αυτό. Είναι ένα έγγραφο ανατολισμού που θέτει τι βάσει. Έλεγε ο κύριο Νίκολσον ότι το έγγραφο είναι πιο, Μάλλον, ε, το έγγραφο πιο σημαντικό για αυτά που δεν λέει παρά για αυτά που λέει. Μα ακριβώ περί αυτού πρόκειται. Η Κομισιόν είπε αυτά που είχε να πει πρότεινε κάποιες κατευθύνσεις, πρότεινε τρεις επιλογές, τρία σενάρια, τα οποία όλα είναι προσυζήτηση. Προτείνουμε επίσης και κάποια μέσα στον πρώτο, στο δεύτερο πυλώνα για τις ε, άμεσες ενισχύσεις, για τις επενδύσεις και για την πολιτική προσέγγιση. Το έγγραφο λοιπόν είναι γενικό, επειδή είναι έγγραφο ανατολισμό όπως είπα, και οι λεπτομέρειες θα έλθουν, όπως ε, είναι φυσικό αυτό, στο πλαίσιο της νομοθετικής δέσμης μέτρων που θα προτείνουμε του χρόνου. Πρέπει να καταλάβετε το εξής. Ίσως να έχουμε και πιο συγκεκριμένες ιδέες. Πριν όμως τις θέσουμε επιτάπητος ε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να σας μπορούμε να σας εξηγήσουμε γιατί προβήκαμε στη μία στην άλλη επιλογή. Και όλα πρέπει να είναι δικαιολογημένα. Και γνωρίζετε επίσης ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε και μελέτες επιπτώσεων Επομένως ε, δεν μπορώ να πω τίποτε παραπάνω. Μπορώ να σας αναφέρω εναλλακτικέ λύσεις, ε, διάφορες προτάσεις και να σας αναφέρω επίσης τις αιτιολογήσεις που δίνουμε. Και αυτό για να γίνει πρέπει να προηγηθούν οι μελέτες επιπτώσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα την απλούστευση, θέλω να πω το εξή. Στόχος μας δεν είναι να περιπλέξουμε τα πράγματα, ούτε να προκαλέσουμε σύγχυση Υπάρχουν ε, οι οικολογικές, οικολογικοί όροι, οικολογική συμμόρφωση και θα υπάρξει προσπάθεια ε, σίγουρα απλούστευση με τους επιτρόπους Νταλή και Ποτότσνικ ε, ήδη είμαι σε επαφή για να δούμε πώς μπορεί αυτό να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο και σαφές, αλλά βέβαια να τηρείται και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τι προτείνουμε λοιπόν, να δώσουμε κίνητρα στους αγρότες για να υιοθετήσουν πρακτικές που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη διάρκεια. Συμφωνώ μαζί σας ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι πρώτα απ' όλα για τους αγρότες, αλλά για τους αγρότες με χρήματα των φορολογουμένων. Δεν θα μου άρεσε λοιπόν μια κατάσταση όπου μέσα σε μια πενταετία ή δεκαετία δεν θα συζητάμε πια καν και θα απαρνηθούμε τελείω την ΚΑΠ γιατί θα πούμε ότι δεν είναι δικαιολογημένη αυτή η δημόσια πολιτική. Δεν προτείνουμε κάτι τέτοιο λοιπόν. Προτείνουμε λοιπόν μέτρα που δεν τα έχουμε βγάλει ω λαγό από το καπέλο μας. Είναι μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν και θέλουμε να τα γενικεύσουμε κάνοντας προτάσεις τι τις σχετικές αγρότε. αγρότες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του, ε, της μικρής γεωργικής ε, του ενεργού αγρότη ή γεωργού, το active farmer, και το capping, τη δέσπιση του ανώτατου όριου. Όλα αυτά θα τα επεξεργαστούμε ακόμη περισσότερο. Τι θα πει ενεργός γεωργός, ενεργός γεωργός. Θα πει δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει τη γη, που παράγει κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ε, περιπτώσεις ε, που τις ενισχύσεις τις λαμβάνουν κάποιοι γεωκτήμονες, που δεν κάνουν τίποτα, που δεν παράγουν απολύτως τίποτε. Θα δούμε ακριβώ τον ορισμό, βέβαια, πώ θα τον διατυπώσουμε. Περί αυτού όμω πρόκειται. Τι θα πει τώρα μικρή γεωργική εκμετάλλευση ίσως να μην αντιλαμβανόμαστε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ε, την ε, έννοια της ε, μικρής γεωργικής εκμετάλλευση στην Πολωνία, σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φιλανδία ή την Ιταλία. Το καταλαβαίνω αυτό και θα πρέπει να εγγύψουμε στον ορισμό. Σίγουρα θα διατυπώσουμε προτάσει. Αυτό που θέλω να πω όμω ότι σημαντική είναι η έννοια, σημαντικό είναι όρο. Το ίδιο είναι και με το κάπινγκ, τη θέσπιση ανώτατου ορίου. Το επίπεδο. Θα πρέπει να κάνουμε αξιολογήσει για να δούμε και αυτό το ανώτατο όριο που ε, προτείνουμε πώς μπορεί να συνάδει και πώς μπορεί να είναι ε, λογικό και να οδηγεί σε ενίσχυση του εισοδήματος. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή ε, τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο, ιστορικές αναφορές στο νέο σύστημα. Υπάρχει μεταβατική περίοδος, αυτή τη στιγμή είναι υπό μελέτη το κατά πόσον θα είναι 2, 3, 5 χρόνια. Πάντω θα υπάρχει μεταβατική περίοδο. Πρέπει να αξιολογήσουμε τα πράγματα και θα σας υποβάλουμε συγκεκριμένη πρόταση για τη μεταβατική αυτή περίοδο. Τώρα για τον κύριο Καπούλα Σάντος που είπατε κάτι για τη μείωση των κερδών ε, και των ωφελών μεταξύ των κρατών μελών. Σας κατανοώ, κατανοώ αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να σας πω το εξής. Για να είναι εφικτή, εφαρμόσιμη και αποδεκτή μεταρρύθμιση θα πρέπει να υπάρξει μια επανεξισορρόπηση η οποία θα είναι αρκετά ανεκτή αν θέλετε για αυτούς οι οποίοι θα δουν να μειώνονται ε, τα εισοδήματά τους. Θα πρέπει λοιπόν να εξεύρουμε ένα σύστημα που θα αποτρέπει μια βίαιη αλλαγή, μια βίαιη μετάβαση για ορισμένους ε, αγρότες. Στόχος μας πάντως είναι αυτή η επανεξισορρόπηση χωρίς όμως ε, επανάσταση γιατί άλλοτε γίνεται αποδεκτή και άλλοτε όχι μια τέτοια επαναστατική αλλαγή. Ο στόχος μας πάντως είναι η σαφής μετεξέλιξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γάλα, θα υπάρξουν προτάσεις οι οποίες ε, θα είναι επιπλέον ε, της μεταρρύθμισης αυτής και ίσως θα προηγηθούν μάλιστα των προτάσεων για τη μεταρρύθμιση. Θα ε, κάνουμε λοιπόν την ανάλυση, θα σας υποβάλουμε την έκθεση πριν λήξουν οι γαλακτοκομικές αποσαστώσεις. Σε ό,τι αφορά τις μειονεκτικές ε, περιοχές, πράγματι θα υπάρχει συγχρηματοδότηση κυρίως ε, και στο δεύτερο πυλώνα, άρα υπάρχει ευελιξία στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν ορισμένες ε, κατηγορίες αγροτών ή συγκεκριμένες περιοχές με συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά όταν θα επανακαθορίσουμε τις βασικές πληρωμές θα θέλαμε στον πρώτο πυλώνα τα κράτη μέλη να μπορούν να επιλέγουν και να δίνουν ένα υψηλότερο βασικό επίπεδο πληρωμών σε αυτές τις μειονεκτικές περιοχές. αυτή είναι η ιδέα μας αυτός είναι ο στόχος μας και στη συνέχεια στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα αφήνουμε το στοιχείο της ευελιξίας που καλύπτεται και αυτό βέβαια από εθνική συγχρηματοδότηση. Να επαναλάβω Euh, euh, ότι το πρασίνισμα αυτό ε, δεν ε, θα έχει αρνητικές ε, συνέπειες σε ό,τι αφορά και τη βιωσιμότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, για τις δημοσιονομικές προοπτικές θα έχουμε με βάση αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν την άνοιξη της προτάσης. Επομένως, τον Ιούλιο θα έχετε την νομοθετική δέσμετρο για την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Υπάρχει μια συνέπεια δηλαδή. Ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα αναλάβουν τις ευθύνες τους όπως τα αναλαμβάνουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε ο προπολογισμό ε, να μπορεί να είναι φιλόδοξο σε σχέση με τους στόχους μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να πούμε ότι ναι, διατηρούμε τον προπολογισμό της κοινή γεωρικής πολιτικής αλλά τελικά ε, προτείνουμε μείωση και ζητούμε από την Κομισιό να χρηματοδοτήσει άλλες πολιτικές. Σε αφορά το παγκόσμιο εμπόριο δεν μπορώ να το συζητήσω εδώ. Είναι ένα θέμα που μπορούμε να το δούμε ξεχωριστά. Δεν είναι ε, μια μεταρρύθμιση την οποία προτείνω σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Για την Ντόχα έχει κάνει την πρότασή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάδει με τις δικές μας προτάσεις για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις τώρα είναι σε εξέλιξη και εγώ δεν φιλοδοξώ να προσαρμόσω την κοινή γεωργική πολιτική σε σχέση με τη μία ή την άλλη διαπραγμάτευση γιατί η κοινή γεωργική πολιτική αφορά πρώτα απ' όλα την ευρώπη και τους ευρωπαίους. δίκτυα ασφαλείας τιμές κατώτατες τιμές ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα των κατώτατων τιμών ήδη με το σύστημα αυτό με το δίκτυο ασφαλείας κατά κάποιον τρόπο περιορίζεται η μείωση των τιμών. Συγκρατούνται οι τιμέ, αλλά στόχος μας είναι να βρούμε και έναν άλλο μηχανισμό που να είναι προσαρμοσμένος στις τρέχουσες αγορές. Τώρα δεν ξέρω ακριβώ αν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το είδος μηχανισμού στην κατάσταση που οι ευρωπαϊκές αγορές θα είναι πιο ανοιχτέ προ τα έξω. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μέσα προστασία. Φυσικά και θα έχουμε. Παραδείγματο χάρη τιμή εισαγωγή για τα απορροκυπευτικά. Υπάρχει. Υπάρχουν φραγμοί δασμολογικοί για το κρέα, για το γάλα, για άλλα προϊόντα. Άρα δεν στερούμεθα πλήρω ε, προστατευτικών μηχανισμών. Απλά πιστεύω ότι στο πλαίσιο τη εσωτερική αγορά θα πρέπει τώρα να εξέρουμε μηχανισμού που θα είναι προσαρμοσμένοι στην τρέχουσα πραγματικότητα. Έξω και δεν διατύπωσα προτάσει που κατά την άποψή μου δεν έχουν τύχει και δεν θα βρουν υποστήριξη στο σημερινό πολιτικό πλαίσιο. Νομίζω ότι λίγο πολύ απάντησα. Eh, Ευχαριστούμε. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, ενάμιση λεπτό αναομιλητή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Ε, η κυρία Λίζα Γέγκελ θα ανοίξει ε, το δεύτερο γύρο στις συζητήσεις μας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω θερμά και τον Επίτροπο. Μας υποβάλλατε ένα έγγραφο το οποίο αποτελεί μια καλή και ευρία βάση εργασίας για την Επιτροπή Γεωργίας. Κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε ήδη ψηφίσει και στην έκθεση Λάιεν, τα οποία αναπτύσσονται περαιτέρω στο έγγραφο. Αυτό σας ευχαριστώ λοιπόν. Και ναι, έχουμε κοινό στόχο να μετεξελίξουμε για την Ευρωπαϊκή Γεωργία την ΚΑΠ. Σκοπό σας επίσης είναι να ορίσετε γιατί χρειαζόμαστε τα κονδύλια αυτά, γιατί χρειαζόμαστε την πολιτική αυτή. Και πολύ έντονα τονίζετε τους περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και την εδαφική ισότητα. Θα ήθελα να τονίσω ευθύ εξ αρχή ότι το μεγαλύτερο καθήκον μας είναι να φροντίσουμε τα 500 εκατομμύρια καταναλωτές τη ευρωπαϊκή Ένωση, να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας και υγιεινά τρόφιμα. Περιγράψατε ευρέω διάφορα στοιχεία, αλλά ε, υπησέρχεστε σε λεπτομέρειες για ένα στοιχείο και ρωτάτε πώς θα πρέπει να το αναπτύξουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Στη σελίδα 6 αναφέρεται και παραθέτω ότι οι διαδικασίες εφαρμογή της ΚΑΠ πρέπει να απλοποιηθούν, θα πρέπει να γίνουν πιο έντονοι οι έλεγχοι και να μειωθούν ε, να μειωθεί το γραφειοκρατικό, το για, τους, ε, για τα άτομα τους δικαιούχους. Ωστόσο, ωστόσο μου δίνει την εντύπωση ότι αυτά τα τρία στοιχεία είναι αντιφατικά. Πώς θα απλοποιήσουμε τις διαδικασίες κάνοντας πιο έντονους ελέγχους και πώς αυτό συνάδει με τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους για τους δικαιούχους. Θεωρώ ότι πρόκειται για αντίφαση, για παράδοξο. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Και να πω ότι η κοινή πολιτική ε, σε ό,τι αφορά τις διμερείς συμβάσεις σχετίζονται αυτά τα δύο γιατί με την Κορέα, με το Μαρόκο, με την Μερικοσούρ, με τον Καναδά έχουμε διμερείς σχέσεις και αν δεν θέσουμε τα δικά μας πρότυπα για πρόσβαση στην αγορά μας θα αποδυναμωθεί εν τέλει και η δική μας αγορά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ Ελίζαμπετ, ο Κώστας. Ε, κυρία ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Νομίζω ότι πολλά ε, έχουν πολύ μεγάλο περιθώριο ερμηνείας στο έγγραφο που σας αναφέρετε. Θα σας ε, δώσω απόλυτο δίκιο. Είναι αναγκαίο να υπάρξει μεγαλύτερη δικαιοσύνη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ισχύει και για όλα τα κράτη-μέλη. Από αυστριακής πλευράς ε, είναι πολύ σημαντικός ο δεύτερος ε, πυλώνας, γιατί εκεί έχουμε το 2 τρίτο, τα 2 τρίτα των ε, ενισχύσεών μας. Και από εκεί χρηματοδοτούνται και οι περιοχές ημιονεκτικές, όπως οι ορεινές περιοχές της Αυστρίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο μέλλον να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τους ε, συναδέλφους που εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τα θέματα τα γραφειοκρατικά. Γιατί ξέρετε αυτά πλήττουν και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβαρύνονται υπερβολικά από τα γραφειοκρατικά και από τους ε, ελέγχους. Λυπάμαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι στην ανακοίνωσή σας ε, δεν ε, γίνεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά για ευαίσθητους τομείς όπως είναι το γάλα. Και σας παρακαλώ, Επιτροπέ, να δώσετε ε, να υπάρξει ήπια προσγείωση σε ό,τι αφορά τους τομείς αυτούς. Γιατί ξέρετε, 4,5 εκατομμύρια είναι άνω των 65 στη Γεωργία και θα έχουν ε, πάρει σύνταξη μέχρι το 2020. Θα πρέπει λοιπόν να θέλουν οι νέοι να παραμείνουν στον ε, αγροτικό κλάδο και αυτό προϋποθέτει ότι θα μπορούν να έχουν ένα σταθερό εισόδημα για το μέλλον. Γκαρσία Πέρεθ, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι φαίνεται να υπάρχει ομόφωνη ε, σχετικά ε, συμφωνία στο πλαίσιο της Επιτροπής του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά γενικά το έγγραφο πρώτα απ' όλα και επίσης συμφωνούμε ότι ανταποκρίνεται στις βασικές προκλήσεις ε, τις οποίες είχαμε και εμείς αναφέρει στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως νομίζω ότι είναι στο σωστό δρόμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις ανησυχίες που εκφράζονται από τον κλάδο αυτή τη στιγμή. Όπως είπαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου, πρέπει να δούμε βέβαια και τα μικρά γράμματα. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα συγκεκριμενοποιήσουμε, πώς θα δώσουμε σάρκα και οστά σε όλα αυτά τα ζητήματα, ώστε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κλάδου. Νομίζω ότι η βασική αρχή για να ανταποκριθούμε στις ε, προκλήσεις και για να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες του κλάδου είναι να είμαστε σε θέση να αγγιηθούμε τα εισοδήματα των Ευρωπαίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Και για να το κάνουμε αυτό συμφωνούμε νομίζω ότι αφενός έχουμε την μέθοδο των άμεσων πληρωμών μέσω του πρώτου πυλώνα που θα δούμε ποια συγκεκριμένη μορφή θα πάρει μέσω των κανονισμών αλλά μπορούμε να το εγγυθούμε και με την καλή λειτουργία της αγοράς. Είναι σημαντικό και θα ήθελα να μας πει ο Επίτροπος πώς θεωρεί ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαπραγματευτική θέση του γεωργού ε, στην αλυσίδα αξίας. Και επίση θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία και η κτηνοτροφία είναι διαφοροποιημένε, ε, είναι πολυπίκυλε. Πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ποικιλότητα αυτή, Πώ μπορούμε να ανταποκριθούμε στι ιδιαιτερότητε ε, του κάθε εδάφου, τη κάθε περιοχή. Παραδείγματο χάρη συγκεκριμένα ζητήματα όπω είναι η κτηνοτροφία του Νότου. Πώ θα τα δούμε, είπατε εσεί ε, πιο βιώσιμη κτηνοτροφία κύριε Επίτροπε. Πώ μπορούμε να διατηρήσουμε την κτηνοτροφία στον Νότο που είναι διαφορετικές οι πραγματικότητε, λόγω ε, λήψη κτλ. και τα λοιπά. Και βέβαια καλό θα είναι να δούμε και κατά περίπτωση ειδικά προβλήματα που ενδέχεται να ανακύπτουν. Ευχαριστώ. E Ο κύριος Τόρφμαν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόρφμαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Πρόεδρε, Επίτροπε, είναι γενικά θετική η στάση μας για την ε, ανακοίνωση αυτή και γίνεται μια έντονη συζήτηση τον τελευταίο, τους τελευταίους μήνες κατά τους οποίες, ε, οποίους ήταν πολύ θετική η ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τις μειονεκτικές περιοχές θεωρώ ότι γίνεται μια σαφής απόπειρα να περάσουμε από τον δεύτερο πυλώνα στον πρώτο. Εγώ είμαι υπέρ των προτάσεων σας αρκεί να υπάρχουν κάποιες εγγύησεις. Και αυτό με φέρνει σε αυτό που σας ζητώ. Θέλω να διευκρινίσετε τις προθέσεις σας, για την πληρωμές για τον πρώτο πυλώνα και σε ό,τι αφορά τις πληρωμές ε, για τον δεύτερο πυλώνα, πώς θεωρείτε ότι θα σταθμιστούν σε ό,τι αφορά τη μελλοντική διαμόρφωση, επίσης σε ό,τι αφορά την περικοπή των πληρωμών. Χαίρομαι που τα αναφέρετε και που προτείνεται σε κάποιες καταστάσεις, οι πληρωμές αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν σε ό,τι αφορά τις ορεινές περιοχές. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Και αν θέλουμε να συνεχίσουμε τις εκτροφές σε ορεινές περιοχές όταν σταματήσουν και οι ποσοστώσεις, θα ε, δυσκολευτούμε πάρα πολύ αν δεν υπάρχουν ειδικέ ε, ρυθμίσεις. Και για το πρόγραμμα λίτε δεν αναφέρεται κατά πόσο θέλετε να συνεχίσει, γιατί είναι καλό πρόγραμμα. Επίσης, θεωρώ ότι είναι σωστό να προχωρήσουμε σε απλούστευση, απλοποίηση των διαδικασιών σε ό,τι αφορά α, τις μικρές επιχειρήσεις και τις μειονεκτικές περιοχές, γιατί θέλουμε τελικά ένα αγροτικό περιβάλλον σωστό. Ο κ. Παπαστάμκος. Κύριε Επίτροπε, καλωσορίζω την σταθερή δέσμευσή σας για μια ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο ζήτημα της δίκαιης κατανομής των ισχύσεων, το οποίο αναδείξατε ως μια από τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές της μελλοντικής ΚΑΠ. Στην ανακοίνωσή σας αναγνωρίζετε σαφώς ότι η ενιαία ενίσχυση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το flat rate δηλαδή, δεν συνιστά λύση, υπογραμμίζω, δεν συνιστά λύση για τη δίκη κατανομή των άμεσων ισχύσεων. Πράγματι υφίστανται ουσιώδεις αποκλήσεις ως προς τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το κόστος παραγωγής, καθώς και στο ποσοστό συμβολής της γεωργίας στην απασχόληση, όπως τόνισε ο κύριος συνάδελφος ο Καπούλα Σάντος, και στην οικονομία στις επιμέρους περιφέρειες. Υφίστανται επίσης φυσικ... σημαντικές φυσικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών και αναφέρομαι μεταξύ άλλων στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, και στις περιβαλλοντικά ευάλωτες περιοχές όπως είναι οι περιοχές του Ευρωπαϊκού Νότου. Θα ήθελατε, θα μπορούσατε να διευκρινίσετε ακόμη περισσότερο, όχι με όρους δέσμευσης, αλλά δικών σας προσωπικών σκέψεων, ποια πιστεύετε κατά τη γνώμη σας ότι πρέπει να είναι η μεταβατική περίοδος, η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων. Και πάλι σε επίπεδο σκέψεων, όχι δεσμεύσεων, ποια αντικειμενικά κριτήρια διερευνά η Κομισιόν για τη δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων. Και κάτι τελευταίο, βεβαίω η Κομισιόν είναι ένα συλλογικό σώμα, είναι το κολέγιουμ των Επιτρόπων, αλλά εσείς ε, κύριε Επίτροπε σας δίνετε η ευκαιρία, η δυνατότητα να κρατήσετε ψηλά τη σημασία, δεχόσαστε πιέσει ασφαλώ από άλλου επιτρόπους που έχουν μια άλλη προσέγγιση στα θέματα, αλλά κρατήστε ψηλά τη σημασία, τη σποδιότητα μιας ισχυρής κοινή αγροτικής πολιτικής, ε, προς το 2020. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σε ευχαριστούμε. Στέφαν Φόλι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Επίτροπο για τις εργασίες των οποίων ηγήθηκε επί σειρά μηνών και των ακροάσεων κυρίως που διοργάνωσε πριν τη θερινή διακοπή. Έτσι να λοιπόν, είπα προσδιορίσαμε στόχους για την κοινή γεωργική πολιτική. Νομίζω ότι αυτό είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας. Δεν θα ευσέλθουμε σε λεπτομέρειες και θα συζητήσουμε τις ανησυχίες και την αγωνία ε, του καθενός και της κάθε χώρας. Θα έρθει η ώρα να τα συζητήσουμε σήμερα. Συζητούμε για τους βασικούς προσανατολισμούς. Ποια, τι είδους κοινή γεωργική πολιτική η Επιτροπή συλλογικά και όχι ο Επίτροπος μας κάνει μια εισήγηση. Και επ' αυτού θα συζητήσουμε και εγώ επ' αυτής της βάσης θα αποτιμήσω, θα αξιολογήσω αυτή την πρόταση. Λοιπόν, η πρόταση ακολουθεί τη σωστή ρότα για πέντε βασικά σημεία που για μένα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Επισητιστική ασφάλεια. Οι Ευρωπαίοι είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε κατοχυρώσει την επιστημιστική μας ασφάλεια μέσα από τη γεωργία μας. Εμείς, εσείς, ε, πρέπει να αναρωτηθούμε αν ισχύει αυτό είναι κέρια σε καταλητική σημασία. Δεύτερον, το θέμα του περιβάλλοντος. Υπάρχει συμμόρφωση με την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε και παραγωγική και βιώσιμη ανάπτυξη. Εσεί ισχυρίζεστε ότι είναι δυνατόν αυτό. Εμείς έχουμε την ίδια συζήτηση στο Κοινοβούλιο και θα συνεχίσουμε να την έχουμε. Πάντως για μένα είναι κέριο το ζήτημα. Τρίτον, το να λάβουμε υπόψη την κοινωνική διάσταση, ε, δηλαδή ενεργός απασχόληση ε, στα πλαίσια της γεωργίας. Ναι, αυτή είναι η σωστή συζήτηση γιατί έτσι θα καλύψουμε και την κοινή γνώμη. Δηλαδή η γεωργία συνδέεται με τους γεωργού, τους ενεργούς γεωργούς. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη καταρτίζοντας την μελλοντική στρατηγική και αυτό το σημείο είναι κέριο κατά τη γνώμη μου. Τελευταίο θετικό στοιχείο ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη της ε, υπαίθρου, την κάλυψη των ε, μειονεκτημάτων κάποιων περιοχών και μερική διατήρηση της σύνδεσης των ενισχύσεων. Για μένα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα θα περάσω στο κομμάτι της ρύθμισης της διαχείρισης των κοινών οργανώσεων αγοράς ε, των μέτρων που συμπεριλαμβάνονται μέσα στο έγγραφό σας. Ε, ε, επ' αυτού, ναι, παραμένετε γενικόλογος. Κάνατε κάποια σχόλια για το δεύτερο πυλώνα. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να διευκρινίσετε διεξοδικότερα αυτά τα στοιχεία. Έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική, θέσατε τη γενική ρότα, αλλά πραγματικά πρέπει να συζητήσουμε διεξοδικότερα διαχείριση των αγορών. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Καλινόφσκι έχει τον λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, το ερώτημα του μέλλοντος της ΚΑΠ είναι ένα από τα βασικότερα ερωτήματα που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αλλαγές που προτείνετε στο εγγραφό σας δεν είναι επαναστατικές. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί δεν πρέπει να υπονομεύσουμε τα επιτέγματα του παρελθόντος σε ό,τι αφορά την ΚΑΠ. Ωστόσο, να τονίσω ότι δεν είναι αρκετά τολμηρέ οι προτάσει σας. Και ένα από τα πιο βασικά στοιχεία τα οποία εσείς, Επίτροπε, θέλετε να καταργήσετε είναι το ιστορικό σύστημα των ε, πληρωμών. Ωστόσο, αυτό αποτελεί, θεωρώ, μία πρόταση. Δεν αναφέρεται, ε, για παράδειγμα, στο έγγραφό σας αναφέρεται κάποια μεταβατική περίοδο για τα παλαιά κράτη-μέλη. Και αυτό τι σημαίνει ότι πέρα από τα 10 χρόνια τα οποία ορίστηκαν στην διάσκεψη της Κοπενχάγης θα προσθεθούν και άλλα 7 χρόνια. Πρόεδρε, πώς θέλετε να συζητήσουμε για 7 ακόμα έτη μεταβατικής περίοδου. Είναι πραγματικά μη κατανοητό αυτό. Σας υποστηρίζω ωστόσο σε ό,τι αφορά την έννοια του ενεργού γεωργού. Νομίζω ότι το 30% των επιδοτήσεων δεν πηγαίνει τελικά στους ε, ενεργούς γεωργούς. Πηγαίνει στους γεωκτήμονες. Άρα θεωρώ ότι είναι σωστή η κατεύθυνση αυτή που προτείνεται. Και χαίρομαι επίσης που θα διατηρηθεί το σύστημα των δύο πυλώνων. Ωστόσο θα πρέπει να είναι πιο ισομερείς οι αναλογίες και θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος βαθμός ευελιξίας. Γιατί οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, οι Γεωργοί διαφέρουν από τους Πολωνούς και από τους Ρουμάνους, για παράδειγμα, Γεωργούς. Πέρα από θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, θα πρέπει να επενδύσουμε στον εξυγχρονισμό του γεωργικού μας συστήματος, προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστικό. Και κάτι ακόμα, η αγορά της ζάχαρης, θα μπορούσατε να πείτε δύο λόγια για αυτή την αγορά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος και ο κύριος Λαβίνια και μετά ο Αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα όπως και οι προλαλήσαντες συνάδελφοί μου να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο που σκιαγράφησε τις γενικές γραμμές της ε, μελλοντικής κοινής γεωργικής πολιτικής συμβαδίζει και με τη συνθήκη της Λισαβόνας και με προηγούμενες προτάσεις της που λέει ότι θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να έχει λόγο. Πράγματι τώρα το μπαλάκι όπως είπαν άλλοι συνάδελφοι είναι στο δικό μας γήπεδο και έχουμε ένα νέο ρόλο να διαδραματίσουμε. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να δώσουμε σάρκα και οστά προτάσεις, να προσθέσουμε λεπτομέρειες διότι θα έχουμε και μια νομοθετική έκθεση η οποία θα καλύπτει πολλούς από τους τομείς που αναφερθήκατε, στους οποίους αναφερθήκατε και τους οποίους εμείς θα εξετάσουμε ως κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτή την γενική σκιαγράφηση πρέπει να πω ότι με ικανοποίησε χάρηκα που άκουσα αυτά που είπατε είπατε για τους πόρους Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να γίνει εδώ είναι να βρεθούν πόροι για χρηματοδότηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη να λυθεί το οικονομικό ζήτημα και βλέπουμε να υπάρχει διελκυστίνδα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Το είδαμε και αυτή τη βδομάδα για τον προπολογισμό του 2011. Υπάρχουν κάποιες χώρες που πραγματικά ε, στόχο έχουν να, να περικόψουν τη συμμετοχή τους στον κοινοτικό προπολογισμό. Είναι λοιπόν ε, σκληρή μάχη που θα πρέπει να δώσουμε για να πετύχουμε και την πολιετή δομή χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν ε, προσβλέπω να ε, υλοποιηθεί αυτή η πολιτική. Θα δούμε τι θα γίνει και κατά το πρώτο εξάμεινο του 2011, παρότι δεν θα έχουμε στις αρχές του έτους την απόφαση για την χρηματοδότηση. Πώ θα μιλήσουμε λοιπόν για τι νομοθετικέ εκθέσει χωρί τη χρηματοδότηση, χωρί να είναι σαφής ο προπολογισμό. Θα λίγο δύσκολο, γιατί θα είμαστε σε ένα κενό, θα είμαστε λίγο μετέωροι, δεν θα ξέρουμε ποιο είναι το πλαίσιο και αυτό θα μας βάλει σε λίγο δύσκολη θέση. Η Αντιπρόεδρος Πάουλσεν, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Επίτροπο. Εγώ θεωρώ πως το έγγραφο είναι σχετικά καλό, γιατί όλες τις πόρτες ανοιχτές τις έχει. και απευθύνεστε στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Γεωργίας και έχετε και όλες τις δύσκολες διαπραγματεύσεις σύντομα με το Συμβούλιο. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Ο Επίτροπος Τσιόλος, κατά τη γνώμη μου, κατάφερε να έχει όλες τις αλλακτικές λύσεις μέσα στο έγγραφο, ακόμη και τις ανέφικτες. Μπράβο! Προσωπικά Χαίρομαι που θα περάσουμε και θα λάβουμε υπόψη την έννοια του ενεργού γεωργού. Προσπάθησα να μάθω ακριβώς πού προσγειώνονται τα λεφτά από την κοινή γεωργική πολιτική. Δηλαδή, γίνεται να έχουμε ένα σωστό κανονικό ορισμό του ενεργού γεωργού. Έχουμε επιχειρήσεις όπως η Nestlé και άλλες που είναι μεγάλοι επιχειρησεις οπως η νεσλε και αλλες που ειναι μεγαλοι δικαιουχοι και αυτοί ανήκουν στη γεωργία, αλλά δεν είναι όμως γεωργοί. Επίσης, οι ενισχύσεις που υπολογίζονται βάσει των ιστορικών δεδομένων χαίρομαι που θα εκλείψουν. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτά τα στοιχεία. Τα Οι φορολογούμενοι, οι καταναλωτές ε, πληρώνουν και πρέπει να συμμετάσχουν στην συζήτηση και στον προβληματισμό. Η οξύτερη κριτική που ακούγεται είναι πρώτον ότι πολλές ενισχύσεις δεν καταλήγουν στους γεωργούς ε, που η κοινή γνώμη συμφωνεί ότι πρέπει να στηρίξουμε ε, πολλές ενισχύσεις πάνε στους μεγάλους ε, γεωκτήμονες, στους εκμισθωτές σε σχέση με τις μικρές εκμεταλλεύσεις που παίρνουν χαμηλότερες ενισχύσεις θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Τσιολώση γιατί η φροντίδα των ζώων επίσης είναι ένα στοιχείο του εγγράφου και τώρα θεωρείται και γίνεται αποδεκτό ότι συνιστά κοινό συμφέρον της Ένωσης και πρέπει να αποτελέσει και κοινή δέσμευση. Σας ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε σε ζητήματα στο μέλλον. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει εντελώ διαφορετική κατανομή ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα. Θα ήθελα επίση να έχουμε μια ε, σαφέστερη αντίληψη περί ε, γεωργίας, πώς ακριβώς θα εξασφαλίσουμε την επιστημιστική ασφάλεια. Αλλά μην ξεχνάτε ότι επί τόπου στα κτήματά μας η γεωργία είναι σημαντική ναι μεν για την επιστημιστική ασφάλεια αλλά έχει και καταλητικό ε, ρόλο για το μέλλον της Ευρώπης, ε, του περιβάλλοντος, την προστασία της βιοποικιλότητας κτλ. Ο πρόεδρος ε, διακόπτει την αντιπρόεδρο Πάουσον, ο κύριος Ράιμερς και Χάλβες ακολουθούν. Ευχαριστώ. Επίτροπε χαίρομαι που ήρθατε εδώ σήμερα. Μιλήσατε και είπατε ότι θέλετε το έγγραφο αυτό να αποτελεί ένα έγγραφο κατεύθυνση. Αλλά επειδή έχει υπάρξει και μία πρώτη έκθεση, θεωρούσαμε ότι αυτό ήταν ε, το έγγραφο κατεύθυνση και θα ήθελα στη συγκεκριμένη φάση να είχαμε πιο πολλέ λεπτομέρειε. Αυτό το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα είναι ότι το έγγραφο αυτό μου μυρίζει γραφειοκρατία, όπω είπαν πολλοί συνάδελφοι, και αυτό δεν θα επιβαρύνει μόνο του γεωργού. θα επιβαρύνει και τα κρατημέλη τους δήμους, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν του ελέγχου στη συνέχεια και όλα αυτά σε μια εποχή που παντού κάνουμε περικοπές. Θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να παρατραβήξουμε το σκηνή στο σημείο αυτό, γιατί αυτό δεν θα είναι πρακτικά εφαρμόσιμο στη γεωργία. Δεν είναι δυνατόν να χρειάζεται ένας γεωργός ε, ε τον ίδιο χρόνο, για την γραφειοκρατική του δουλειά όσο χρειάζεται για τη δουλειά του ε, στις αγρούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους 16 εκπροσώπους οργανώσεων παραγωγών από τις Ασόρες που βρίσκονται εδώ για να ε, συμμετάσχουν στο διάλογο περί μεταρρύθμισης. Τρεις είναι οι βασικές προκλήσεις. Ε, βιωσιμότητα, οικονομική και περιβαλλοντική σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχουμε ε, κατοχυρωμένη την επιστημιστική ασφάλεια με υψηλές ρυθμιστικές απαιτήσεις για να έχουμε ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές και επίση η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να είναι κοινή πολιτική με κοινού κανόνε ε, για να στηρίξει τη γεωργία και τα εδάφη σε ολόκληρη την επικράτεια τη Ένωση. Θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ με την οικονομική βιωσιμότητα μια γεωργία που θα καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια τη Ένωση. Είμαστε στα 2.000 χιλιόμετρα από τη γυραιά Ήπειρο στι Ασόρε και έχουμε ιδιάζουσε κλιματολογικέ και περιβαλλοντικέ συνθήκε. Έχουμε ελεγχόμενη παραγωγή, έχουμε μεγάλη παραγωγή γάλακτο που αντιστοιχεί στο 30% και άνω τη παραγωγή Πορτογαλία. Σε ένα ελάχιστο ποσοστό, ε, με ένα ελάχιστο πληθυσμό. Παρόλα αυτά είμαστε βασική εξαγωγή και για όσου ασχολούνται με τη γαλακτοπαραγωγή γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το θέμα για τι Αζόρε. Πώ θα εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα όταν εκλείψουν οι γαλακτοκομικέ ποσοστώσει. Ε, ήδη πρέπει να διασχίσουμε 2.000 χιλιόμετρα για να πάμε στι αγορέ. Πώ θα συμμετάσχουμε εμεί στο εμπόριο. Θα, επίσης ε, θέλουμε δικαιότερε συνθήκε για να ανταγωνιστούμε με του συναδέλφου από την Ήπειρο που βρίσκονται δίπλα στι αγορέ. Πώ θα ανταγωνιστούμε όταν πρέπει να διασχίσουμε αυτή την τεράστια απόσταση στη θάλασσα και πώς ε, ε, ενώ πρέπει να αποθηκεύουμε αυτά τα ευπαθή γαλακτοκομικά προϊόντα θα πρέπει να καθησυχάσετε επίτροπε τους γεωργούς και να εξασφαλίσει την επίτευξη αυτού του στόχου δηλαδή της ε, αλληλέγγυας και κοινή για όλους γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η επιλογή του να γίνει συζήτηση εδώ στο ημικύκλιο μας δείχνει πολύ καλά ότι δεν είναι ένα θέμα του παρελθόντος η γεωργία, αλλά είναι ένα θέμα του μέλλοντος και ότι αφορά ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνία. Και εσείς στην ανακοίνωσή σας μιλήσατε ε, για την προτεραιότητα ε, που αντιπροσωπεύει η παραγωγή τροφίμων. Και εμείς λοιπόν θέλουμε ποιοτικά και υγιή τρόφιμα θέλω πραγματικά να αποτίσω φόρο τιμή σε εσά, κύριε Επίτροπε, γιατί το έγγραφο το οποίο μα ε, παρουσιάσατε σήμερα δεν είναι δικό σα έγγραφο, είναι έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τι προηγούμενε μέρε και εβδομάδε καταφέρατε έναν έναν όλου του ομολόγου σα να του πείσετε, να του εισπυρώσετε στο πλευρό σα. Βασιζόμενο σε μεγάλο βαθμό και στην έκθεση την οποία είχε εγκρίνει το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο. Επομένω. Ε, βλέπουμε ότι σε σχέση με την πολιτική των 15 τελευταίων ετών υπάρχουν τομές. Δεν είναι μόνο η γεωργία ε, ο τομέας. Ε, θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια και το νομοθετικό κείμενο, αλλά είμαστε διαθέσιμοι, το είπαμε και το επαναλάβαμε, έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες σας για να έχουμε ένα πολύ καλό έγγραφο για τη δύσκολη περίοδο διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσει. Βέβαια, είναι προφανές ότι έχουν ανασταλεί οι διαπραγματεύσεις λόγω των δημοσιονομικών συζητήσεων και έχουμε και το δίκαιο ανταγωνισμού που πρέπει να συζητήσουμε. Περιμένουμε λοιπόν τι εξέλιξη θα υπάρξουν στα δύο αυτά μέτωπα. Το έγγραφό σας νομίζω ότι αποσιωπά αρκετά το θέμα της διαγενειακής ανανέωσης που νομίζω είναι μια από τις μελλοντικές προκλήσεις, όπως επίσης και το ζήτημα της επανεξισορρόπησης των παραγωγών στην Ευρώπη, λόγω της ανταγωνιστικότητας που θα έχει η γεωργία των χρόνων της κεντρικής Ευρώπης. Προτείνεται επίσης ένα πρασίνισμα που ίσως είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική, αλλά θα δούμε και τι θα γίνει με κάποια μέτρα ενσωμάτωσης. Αν θέλουμε να βάλουμε ακόμα ένα βάρος στις πλάτες των αγροτών, δεν θα μπορέσουμε να σας ακολουθήσουμε σε αυτό το δρόμο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα την πρόεδρο Ζωζέ Μποβέ. Ευχαριστώ και εγώ καταρχάς να ευχαριστώ με τη σειρά μου τον Επίτροπο Ντάσιαν Τσιόλο. Ε, πρώτα απ' όλα για τον τρόπο με τον οποίο εκπώνησε την έκθεση αυτή, διότι είναι η πρώτη φορά που μια τόσο σημαντική έκθεση, ένα έγγραφο μεταρρυθμιστικό, ε, εκπονείται μετά από ευρείες διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, με επαγγελματικές γεωργικές ε, οργανώσεις και με το σύνολο όλων όσων ήθελαν να συμμετάσχουν. Αυτό έγινε τον Ιούλιο, πριν από κάποιους μήνες δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που το Κοινοβούλιο, τα κράτη και η κοινωνία των πολιτών ε, μαζί επεξεργάζονται ένα πρόγραμμα και θέλω να ευχαριστήσω τον Επιτρόπο για αυτό. Υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα που λέγεται, λέγονται στο έγγραφο. Δεν θέλω να απαριθμίσω κι εγώ με τη σειρά μου τα θετικά στοιχεία, απασχόληση, θέση ψανοτατορίου κτλ. Θέλω όμως να αναγνωρίσω ε, τις τρεις ε, λειτουργίες, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική που έχει το λειτουργήμα του αγρότη. Τι προσφέρει λοιπόν ε, η Πέθρος, τι προσφέρει η Γεωργία στις περιοχές. Όλη αυτή, αυτή η προσφορά και αυτή η σχέση δείχνει ότι αν δεν γίνει σεβαστή η γη, το νερό, η βιοπικιλότητα, δεν υπάρχει γεωργία. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ισορροπία μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας, βιοπικιλότητας. Και όλα αυτά είναι στο επίκεντρο αυτού του εγγράφου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάτι πάντως το οποίο είναι λίγο ακόμη ακαθόριστο είναι ο έλεγχος των παραγωγών. Της παραγωγής δηλαδή. Γιατί πώς, ε, αν δεν ελέγξουμε τους όγκους παραγωγής, ε, τι θα κάνουμε το θέμα της ε, προσφοράς και της ζήτησης. Και αυτό σχετίστηκε με το κόστος παραγωγής. Και κάτι άλλο είναι η σχέση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας με τον υπόλοιπο κόσμο, που δεν είναι ακόμα ε, πολύ καλά καθορισμένο στην έκθεση. Είπατε ότι είναι μια γενική έκθεση, είναι πράγμα, το καταλαβαίνω αυτό. Ε, και ζούμε ιστορικές στιγμές, συμφωνώ. Ασχολούμαι με την ε, γεωργία από την εποχή Μάνσχολτ, επιτρόπου Μάνσχολτ. Από τότε η γεωργία, μάλλον τότε οι αγρότες είχαν πάψει ίσως να έχουν μέλλον, τώρα πλέον έχουν πάλι μέλλον. Και θέλω εκ μέρους των αγροτών να σας ευχαριστήσω και εσάς κύριε Επίτροπη για αυτό. Ευχαριστώ Ζωζέ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο μόνο σε τακτικά μέλη της Επιτροπής. Ε, κύριος Ντότζ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο. από, πολλοί από τους ψηφοφόρους μου θα χαρούν σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση που ακολουθεί το έγγραφο της Επιτροπής και στην ε, Βόρεια Ιρλανδία θα λέγαμε, όπως είπε και ο συνάδελφος Ντές, ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στην αρχή εξηγήσατε ότι θα πρέπει να νομιμοποιήσουμε την αγροτική πολιτική. Και Μία μορφή νομιμοποίηση είναι η ανάγκη επισυντηστική ασφάλεια στην Ευρώπη. Όχι μόνο επαρκής ε, ποσότητα τροφίμων, αλλά και ασφαλών τροφίμων με ανιχνεσιμότητα. Υποστηρίζουμε το σύστημα των δύο πυλώνων και ξέρω ότι θα είναι δύσκολη η συζήτηση για τον προπολογισμό του επόμενου μήνες. Είναι σημαντικό όμω ο κλάδο να γνωρίζει πώ πρόκειται να γίνει η κατανομή των κονδυλίων και τι θα γίνει σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές διαφορές. Θα θέλαμε να ξέρουμε στη Βόρεια Ιρλανδία πώς ε, ορίζεται τον εργό γεωργό και τον ε, ισολογισμό που θα πρέπει να κάνει, την ισορροπία που θα πρέπει να γίνει μεταξύ των πρακτικών ε, και της θεωρίας. Καλωσορίζουμε λοιπόν την θεωρία σας, την, την προσοχή που δίνετε στα εργαλεία της αγοράς σε ό,τι αφορά και την ανταπόκριση στις ε, κρίσεις και η τρέχουσα κρίση προκλήθηκε στην τομέα του γάλακτος, προκλήθηκε από την καθυστερημένη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ε, τελευταία ολομέλεια κοιτάξαμε και θέματα που αφορούν ε, τις εκτροφές. Τέλος, θα θέλαμε να πούμε ότι δεν είναι σωστό να αυξηθεί ο γραφειοκρατικός, η γραφειοκρατική επιβάρυνση στον κλάδο αυτό αντί για την νομιμότητα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. και μετά Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν έχω εγώ το λόγο. Stop. Σταματήσω. Όχι, εντάξει κύριε Μαγκίνε, παρακαλώ. Χαίρομαι, χαίρομαι που υπάρχουν και κύριοι. Gentlemen. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα να πάμε λίγο πιο πριν, γιατί με απασχόλησαν κάποια εισαγωγικά σχόλια. Μην μας αφήσετε να ζητάμε συγγνώμη στην Επιτροπή Γεωργίας για την γεωργική πολιτική, γιατί πολλά άκουσα περί ε, νομιμοποίησης και δικαιολόγησης και όλα αυτά μου ακούγονται σαν απολογία. Ας μην το κάνουμε αυτό. Η γεωργική πολιτική έχει αποφέρει μεγάλη ποσότητα ποιοτικών τροφίμων στους καταναλωτές. Αυτό είναι η δικαιολογία. Δεν χρειάζεται και τίποτε άλλο. Ίσως χρειάζεται κάποια δικαιολόγηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό όμως δεν μας αφορά εμάς. Επίσης να πω ότι χτες και αυτό δεν αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, ο ΟΗΕ προειδοποίησε την παγκόσμια κοινότητα ότι επίκειται νέα επισκεπτική κρίση. Και πού πηγαίνουμε λοιπόν με την ε, γεωργική πολιτική για να δείξουμε προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να δούμε το καθεστώς που μεταρρυθμίσαμε για τη ζάχαρη πρόσφατα. Έχουμε τώρα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη ζάχαρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μεγάλες εταιρείε δεν έχουν την ποσότητα που χρειάζεται. Η Ιρλανδική βιομηχανία ζάχαρης ε, έκλεισε τελείως. Ολοσχερός καταστράφηκε. Να προσέχουμε λοιπόν τι κάνουμε σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα, την πράσινη διαμόρφωση της ε, γεωργικής πολιτικής. Μία λέξη έχω να πω. Ένα είναι μόνο χειρότερο από τη γραφειοκρατία. Είναι το πρασίνισμα της ε, γραφειοκρατίας. Γιατί εδώ έχουμε και γραφειοκρατία και μάλλον έχουμε γραφειοκρατία και για τις περιβαλλοντικές πτυχές και αυτά θα πνίξουν τους γεωργούς. Καλώ ορίζω τις δεσμεύσεις για τα μέτρα της αγοράς και αυτά χρειάζονται γιατί όταν χρειάζονται όταν υπάρχει αστάθεια στην αγορά χρειαζόμαστε τέτοια μέτρα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν. Για τον προπολογισμό, ξέρετε ότι Υπάρχουν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά τον ε, προπολογισμό για τον 2011. Να πω ότι οι διαπραγματεύσει, ω συγκήτρια, οι διαπραγματεύσει δεν πηγαίνουν καλά σε ό,τι αφορά την περίοδο μετά από το 2013. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να απολογούμαστε. Θα πρέπει να ζητούμε τον απόλυτα απαραίτητο προπολογισμό. Το μεγάλο θέμα για, τον Γεωργο, για τους γεωργούς γιατί έχω συναντηθεί με πολλούς εξ αυτών στην Ιρλανδία, είναι ότι δεν βγάζουν αρκετά χρήματα από τη γεωργία και αυτό θα πρέπει να αλλάξει η γεωργική πολιτική. Θα πρέπει να εγγυηθεί ένα εισόδημα αξιοπρεπές για τους γεωργούς. Και καλωσορίζω, Πρόεδρε, την σελίδα 10 της έκθεσής σας, αλλά... Πρόκειται για ένα τελικό σχόλιο, δύο παραγράφων σε ό,τι αφορά την τροφική αλυσίδα. Και αναφέρεται ότι Αλλού υπάρχουν περικοπές, αλλού υπάρχουν ε, αυξήσεις των τιμών, αλλά δεν έχετε συγκεκριμένες προτάσεις. Και επειδή περίμενα πάρα πολύ και επειδή έχει θερμανθεί η συζήτηση, θα ήθελα να υπεραμεινθούμε της πολιτικής μας και να προσέξουμε σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που προτείνουμε. Πρόεδρος Βασεβόσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ε, κάνετε αυτή την παρουσίαση σε μια δυσχερέστατη στιγμή γιατί επισκιάζεται αυτή η συζήτηση από μια άλλη πολύ δύσκολη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ο, ο Πολωνός συνάδελφός σας από την Επιτροπή δυστυχώς είπε ότι χρειάζονται περικοπές στην κοινή γεωρική πολιτική. Ακόμη και αν ισχύει αυτό, δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουν τελικά ουσιαστικά τα προγράμματά μας. Εγώ νομίζω ελπίζω ότι θα βρεθεί μια λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά δεν θα επικρατήσει αυτή η πρόταση περί περικοπής κονδυλίων. Έχετε την αμέριστη υποστήριξή μας ε, για την ε, με νέα μεταρρύθμιση. Συμφωνούμε ότι η επιστημιστική ασφάλεια είναι το πλέον σημαντικό θέμα. Φυσικά πρέπει να υπάρχει ε, ισότιμη κατανομή, προστασία του περιβάλλοντος, όλα αυτά που προαναφέρεται, αλλά όπως και η κυρία Μαγκίνες, εγώ πιστεύω ότι κρύβεται ο διάβολος μέσα στις λεπτομέρειες και ε, για ποιες λεπτομέρειες μιλώ για τον ορισμό του ενεργού γεωργού. Δεν έχουμε ε, σαφείς ε, ακριβείς ορισμούς. Ο γενικότερος όμως προσανατολισμός της πρότασής σας μας ικανοποιεί. Δεν μπορώ να φανταστώ μετά τη μεταρρύθμιση να έχουμε πάλι δύο Ευρώπες, την παλιά και την καινούρια χρειαζόμαστε μια ισορροπή στην Ευρώπη. Η βασική αρχή λοιπόν θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη, η ισονομία. Θα ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκουτιέρες. Muchas gracias. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για το έγγραφο που μας παρουσίασε, διότι είναι και ένα συνεπές, ένα συνεκτικό έγγραφο. Κάποιες φορές ε, είχαν γίνει κάποιες ε, διαρροές ε, μάλλον οι τελικά όμως δεν επιβεβαιώνονται και είναι πάρα πολύ καλό το, το έγγραφο αυτό. Συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι αυτό που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι οι έννοιες, η θεωρία. Συμφωνούμε σε αυτό. Θέλω όμως να αναφέρουμε τις τέσσερις αρχές επί των οποίων συμφωνήσαμε και στο έγγραφο για την ε, ΚΑΠ μετά το 2013. Δηλαδή βιώσιμη περιβαλλοντικά, δικαιότερη, ισχυρότερη και κοινωνικότερη κοινή γεωργική πολιτική. Και νομίζω ότι οι δύο πρώτες ε, αρχές ε, αναφέρονται, καλύπτονται αρκετά ε, στο έγγραφο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις δύο τελευταίες, δηλαδή τη μεγαλύτερη ισχύ και το μεγαλύτερο κοινωνικό χαρακτήρα της κοινή γεωργικής πολιτικής, υπολείπεται το έγγραφο αυτό. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναλάβει την ε, ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγυηθεί μια ισχυρότερη ΚΑΠΑ, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να έχει και η πολιτική αυτή ένα μέλλον. Ένα μέλλον ε, τουλάχιστον ε, άμεσα αρκετά ικανοποιητικό. Επίσης είπατε ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη νομιμότητα στην κοινή πολιτική. Έχει να κάνει κυρίως με τις ε, έννοιες που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ΚΑΠ. Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, των άμεσων ενισχύσεων με τη δημιουργία απασχόλησης δεν υπάρχουν πολλές, ε, πολλές, δεν υπάρχει μεγάλη σχέση. Πρέπει όμως ε, ιδίω οι νέοι, ιδίω οι γυναίκες να ληφθούν υπόψη, γιατί είναι το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πώς μπορούμε λοιπόν να, να συσχετίσουμε την πολιτική αυτή με την παρουσία μεγαλύτερου αριθμού ε, γυναικών και νέων στην Ήπεθρο. Και ένα απλό ερώτημα. Συμπεριλαμβάνουμε καινοτόμα μέτρα για την αύξηση του αγροτικού πληθυσμού, των γυναικών, των νέων. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για την πολιτική αυτή, ιδίως για το χρονικό μετά το 2013. Σικυριέσκη. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να είχατε συμπεριλάβει περισσότερα στοιχεία στην ανακοίνωση τη δεδομένη κατάσταση. Γνωρίζουμε τι έγινε στι διαπραγματεύσει με τον προπολογισμό. Ε, βιώνουμε μια περίοδο οικονομικής κρίσης αλλά φυσικά πρέπει να καλύψουμε τις ιδιαιτερότητες ε, της γεωργίας. Έχουμε δαπανίσει δισεκατομμύρια προς διάσωση των χρηματοπιστωτικών αγορών και τώρα συζητούμε για τη γεωργία που είναι κέρια σημασία. Με ομιλούμε για τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Συζητούμε τι θα συνέβαινε αν δεν είχαμε κοινή γεωργική πολιτική. Και παρόλα αυτά ε, κάνουμε, ε, περικόπτουμε τις ε, δαπάνες Όμως χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία και αυτό οφείλουμε να το αναφέρουμε ρητά. Χρειαζόμαστε διαφοροποιημένη παραγωγή. Φυσικά υπάρχει διαφοροποίηση στην παραγωγή δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ενιαία προσέγγιση για όλους τους τομείς ε, της γεωργίας. Χρειαζόμαστε διαφοροποιημένα μέσα στήριξης ε, για τη γεωργία. Χρειαζόμαστε παρέμβαση ε, υποδεδομένων συνθήκων. Επίσης, ε, πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίξουμε το εισόδημα των ε, μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γιατί απορροφούν το πλεόνασμα της αγοράς εργασίας, προσφέρουν θέσεις απασχόλησης ε, στις εκμεταλλεύσεις. Θα μπορούσατε επίσης να μας μιλήσετε για αυτό το ανώτατο όριο των πληρωμών. Πώς θα, θα περιοριστούν οι πληρωμές, θα υπάρχει ανώτατο όριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας κάθε χρόνο. Ε, παρουσιάζει διλήμματα ε, ε, η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής αλλά το βασικό σου χαρακτηριστικό είναι ότι χαρακτηρίζεται από άνηση μεταχείριση για πολλούς από τους γεωργίους της Ένωσης. Θα ήθελα να σας επενέσω πάντως γιατί δείξατε εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας και προετοιμάζοντας την παρούσα μεταρρύθμιση έχετε τη σωστή βούληση, έχετε προσδιορίσει με σαφήνεια τους στόχους Τώρα βέβαια για τα συγκεκριμένα μέσα υλοποίηση γνωρίζουμε ότι δεν θα τα επιβάλλεται και αυτό το τελευταίο σημείο ε, απασχολεί όλους ιδιαίτερως τους βουλευτές. Ας περάσω στι ερωτήσεις. Για τον πρώτο πυλώνα, ε, νομίζω ότι βάσει του οράματος αυτή η πολυαναμενόμενη ευελιξία ε, συμπεριλαμβάνεται στην ανακοίνωση αλλά δεν θα πρέπει να απλήξει την ανταγωνιστικότητα της ε, ε γεωργίας. Ε, επίσης ε, υπάρχει μια ανισορροπία ανάμεσα στα παλιά και στα νέα κράτη-μέλη και ανάμεσα στα, στις εκμεταλλεύσεις διαφορετικού μεγέθους και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι δυνατότητες για τα νέα κράτη-μέλη ώστε να καταργηθεί αυτή η ανισότητα στις άμεσες ενισχύσεις μέχρι το 2013 και όχι το 2016 όπως προβλέπετε για κάποιες ε, χώρες, για τα διάφορα τώρα κριτήρια επί των οποίων θα υπολογίσετε τις νέες ενισχύσεις, ποια θα είναι η νέα βάση αναφοράς που θα χρησιμοποιήσετε. Επίσης με ενδιαφέρει η άποψή σας ε, για τις δυνατότητες υπολογισμού των ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ, χρησιμοποιώντας κριτήρια που θα βασίζουν στις περιφερειακές ιδιαιτερότητες ε, και στις συγκεκριμένες ποικιλίε που καλλιεργούνται. Ο κύριος Δελάς... Κύριε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που βρίσκεται εδώ σήμερα και που προτίθεται να ξεκινήσει αυτή τη μακρά συζήτηση. Αύριο θα παραβρεθεί στην Ολλανδία για να μιλήσει και με νεαρούς γεωργούς και ελπίζω να καταστεί πιο σαφέ αυτό που προτείνει. Και επειδή οι νέοι γεωργοί είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ανταπεξέλθουν με το νέο αυτό σύστημα, θα ήθελα να αναφερθώ στους επένους ε, του Επιτρόπου για τους δύο πυλώνες. Αλλά να πω το εξή για τον πρώτο πυλώνα παραμένετε πάρα πολύ ασαφείς παρά τις ερωτήσεις που, ζητούν, που θέτουν οι συνάδελφοι. Για τον δεύτερο πυλώνα έχετε περιλάβει ένα πολύ μεγάλο κατάλογο. Ξέρετε, θα έρθει και ο Άι Βασίλη σε λίγο και τα παιδιά φτιάχνουν καταλόγους και λίστες με αυτά που θέλουν. Ε, τι να σας πω, αυτό μου θυμίζει και ο κατάλογος που έχετε φτιάξει για όλα αυτά που ζητάτε από το δεύτερο πυλώνα, ε, ανταγωνιστικότητα, ε, περιβάλλον και ούτω καθεξής και πολύ συχνά όλα αυτά είναι και αντιφατικά με αυτά που λέτε για τον πρώτο πυλώνα και όλη αυτή η ποικιλία των στόχων που ζητάτε από το δεύτερο πυλώνα, γιατί να μην μπουν κάποια στοιχεία και στο πρώτο πυλώνα, αντί να επιμείνουμε σε αυτά τα συστήματα πολλαπλής συμμόρφωσης. Και επίση όλα αυτά θα πρέπει να συγχρηματοδοτηθούν, γιατί ξέρετε ότι κάποιε χώρε ούτε θα το θέλουν, ούτε θα το μπορούν να το κάνουν αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν, να υπάρχουν κοινοί όροι, να υπάρχουν ίσε συνθήκε. Ο Μαξέρ ήταν ο μεγαλύτερο μεταρρυθμιστή, αλλά το όραμά του ήταν κοινό και ευρωπαϊκό. Και εγώ πολύ φοβάμαι, κοιτώντα πόσο ασαφεί είναι οι ιδέες, ότι το δικό σα όνομα θα περάσει στην ιστορία ως το όνομα εκείνου που ε, έχασε τον κοινοτικό χαρακτήρα και που το άφησε να επιστρέψει το όλο ζήτημα στα εθνικά κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να διαφυλάξουμε τον κοινοτικό ευρωπαϊκό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σας ευχαριστούμε κυρία Πατράου Νέβες τώρα. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, θα ήθελα να σας χαιρετήσω, να χαιρετήσω το σημερινό έγγραφο που έτυχε τη συνένεση του Σώματος των Επιτρόπων όπως ακούσαμε νωρίτερα και σας ευχαριστούμε για το ανοιχτό πνεύμα, το πνεύμα συνεργασίας που σας διακρίνει ε, και θα ενόψει αυτού του διαλόγου που θα γίνει για τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ήθελα να χαιρετήσω τους εκπροσώπους των γεωργών της Πορτογαλίας και ιδιαίτερα των ε, παραγωγών από τις Αζόρες. Όπως είπαμε νωρίτερα, ε, θα επικεντρωθούμε στα ρεξικέλευτα στοιχεία αυτής της ε, ανακοίνωσης ε, σε σχέση με προηγούμενες εκδοχές του εγγράφου από τη υπηρεσιακή διαβούλευση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ασκείται πίεση όχι για τους γενικότερους προσανατολισμούς, αλλά για τα ειδικότερα στοιχεία. Λοιπόν, ε, μιλάμε για διαφοροποίηση των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Αυτό το θέμα με ανησυχεί και ρωτώ. Στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων θα αποδοθεί προτεραιότητα στις δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό αναφέρεται στο έγγραφο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις λοιπόν ε, στα πλαίσια του προγράμματος Natura Natura 2000 και την ενίσχυση των υφισταμένων ε, ε, περιβαλλοντικών μηχανισμών προς ενίσχυση αυτών των δράσεων και τι θα γίνει πέρα από αυτή την γνωστή πολλαπλή συμμόρφωση, θα προκύψουν νέε δράσει και πώ θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα νέα μέτρα, μόνο μέσα από την κοινή γεωργική πολιτική. Αυτό θα ήταν λίγο ανησυχητικό αν ίσχυε. Τώρα περνώ στη δεύτερη πτυχή. Για τι ειδικέ ενισχύσει, για τι μειονεκτούσε περιοχέ. Αναφέρεται ότι ένα μικρό τμήμα του πακέτου ε, μέτρων μπορεί να περάσει από το δεύτερο στον πρώτο πυλώνα. Θεωρείται ότι αυτή η μικρή αλλαγή καλύπτει τις ανάγκες της γεωργίας ε, στις μειονεκτικές ε, περιοχές ε, στα πλαίσια των αυστηρών μέτρων λιτότητας που αντιμετωπίζουν κυβερνήσεις πολλών κρατών μελών. Επίσης θα εξαγγείλεται νέο σύστημα λοιπόν των, της ενίσχυσης για, για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Θα έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο άμεσα ενίσχυσης όπως είδαμε σε προηγούμενες εκδοχές του εγγράφου διπεροσιακή διαβούλευση. Επίση ακούσαμε ότι υπάρχει και η αξιολόγηση του αντικτύπου για την πάυση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Μα πότε θα γίνει αυτή η αξιολόγηση ταχύτητα γιατί οι αποφάσει που έχουν ελαφθεί στο παρελθόν μπορεί να είναι δεδειγμένε δεδομένε τη τωρινή κατάσταση και να πρέπει να αναθεωρηθούν. Σα ευχαριστούμε κυρία Βατρανέβε, ο κύριο Αγιούζο και μετά η κυρία Λούλινγκ. Κύριε Γιούς, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε που μας παρουσιάσατε εδώ αυτό το έγγραφο. Ένα έγγραφο που κάνει μια καλή διάγνωση καταρχάς της κατάστασης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Δεν προτείνει όμως λύσεις ε, στη συνέχεια για όλα αυτά τα προβλήματα. Του λείπει το, το δημοσιονομικό στοιχείο. Δεν έχει μια ξεκάθαρη αναφορά στην κατανομή των πόρων τι θα γίνει με την ομαλή μετάβαση για να μην έχουμε δραματικές προσαρμογές όπως λεγόταν στο πρώτο έγγραφο η διαχείριση των αγορών δεν είναι αποτελεσματική, δεν προβλέπονται αποτελεσματικά μέσα για να καταπολεμηθεί η διακύμανση των τιμών και η ερδοσκοπία. Ούτε προβλέπεται κάποιο ταμείο διαχείριση κρίσεων όπω είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει πρόταση για τη βελτίωση τη διαπραγματευτική δύναμη των γεωργών και κτηνοτρόφων στο πλαίσιο τη ε, διατροφική αλυσίδα, παρά το γεγονό ότι αναγνωρίζονται οι απώλειε που υφίστανται σε αυτή την αλυσίδα δεν αναγνωρίζεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η καλύτερη αγροτική ανάπτυξη είναι μια παραγωγική γεωργία. Αγρότες που θα έχουν αποδοτικά εισοδήματα από τη γεωργία. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά η πράσινη γεωργία ε, έχει να κάνει και με κάποιους κανόνες και με κάποιες ε, δαπάνες που έχουν ως αποτέλεσμα τα προϊόντα των Ευρωπαίων αγροτών να μην είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τα προϊόντα εισαγωγής. Υπάρχουν μηχανισμοί που σίγουρα μπορούν να βελτιωθούν. Δεν υπάρχει όμω έλεγχο των μηχανισμών αυτών. Άρα δεν τηρούνται και αυτά τα οποία προβλέπονται. Τέλο, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σα παρακαλέσω να μα ορίσετε ξεκάθαρα τι θα πει εν ενεργεία αγρότη, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο. Και επίση, αντί να μιλάμε για εν ενεργεία αγρότη, καλό θα ήταν να μιλάγαμε για ενεργή παράγουσα γεωργική εκμετάλλευση, διότι η καλλιέργεια της γης είναι κάτι πολύ ευρύ και καλό θα ήταν να μιλάμε για γεωργικές εκμετάλλευσεις και όχι για αγρότες. Τέλος κύριε Επίτροπε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις διαπραγματεύσεις, ιδίως για να υπερασπιστείτε και ένα φιλόδοξο προπολογισμό που ουσιαστικά αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε με την κυρία Λούλινγκ ως τελευταία ομιλήτρια. President. Πρόεδρε, είναι τέλειο που είμαι τελευταία, γιατί αρέσει αυτό στις γυναίκες να έχουν τον τελευταίο λόγο, το ξέρετε αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Ε, ε, ε σας επένεσαν πάρα πολύ οι συνάδελφοι. Πολλές φιλοφρονήσεις σας έκαναν και επειδή εγώ δεν πρόλαβα να εξετάσω εντελεχώς την ανακοίνωσή σας καθότι έφτασε γύρω στο, στις 12 και εγώ είχα λυμμένες υποχρεώσεις. Δεν θα ήθελα να ε, σας επενέσω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Γιατί σας το είπα, δεν πρόλαβα ε, να εξετάσω διεξοδικά την πρόταση. Και όπως πολύ ωραία τα είπε ο κύριος Ντέσε, ε, ο συντονιστής μας και ο εισηγητής μας, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Άρα προσοχή. Πάντως, όπως και άλλοι, νομίζω με ασφάλεια μπορώ να πω ότι στο σωστό δρόμο είστε. Ε, για μένα τι έχει ιδιαίτερη σημασία. Να μεταφέρουμε το μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις τρίτες χώρες πως ε, δικαιούμεθα να έχουμε μία κοινή γεωργική πολιτική και να την χρηματοδοτούμε και να τη διαμορφώνουμε κατά το δοκούν, εξασφαλίζοντας έτσι ότι θα υπάρχουν γεωργοί σε όλες τις περιοχές, ακόμη και στις περισσότερο μειονεκτικές περιοχές όπως η δική μου και ότι αυτοί οι γεωργοί θα δικαιούνται ένα εισόδημα δίκαιο και συγκρίσιμο με άλλες ε, παρεμφερείς πληθυσμιακές ομάδες της περιοχής τους. Δεν ευθύνεται η κοινή γεωργική πολιτική για όλα τα δεινά, έτσι, για τις τρίτες χώρες, για τις χώρες ΑΚΕ που κρίνουν ότι λόγω της κοινή γεωργικής πολιτικής έχουν ε, πέσει στη φτώχεια. Όχι, δεν ισχύει αυτό και πρέπει να του εξηγήσουμε. Εγώ πάντοτε, πάντοτε του το εξηγώ και στο Γερολάτ τώρα του το ξαναεξήγησα. Μα αφού δικαιούμαστε στην Ευρώπη να έχουμε μία ε, να έχουμε γεωργική ε, παραγωγή σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Λοιπόν, τώρα το ε, δίκαιο εισόδημα, δυστυχώς κύριε Αντιπρόεδρε, δεν εξασφαλίζεται από τις τιμές των τροφίμων στις χώρες μας οι καταναλωτές. Είναι οι πλέον ευνοούμενοι από αυτό το χαμηλότατο επίπεδο τιμών που δεν αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής και ιδού, ο λόγος για τον οποίο δικαιολογούνται οι άμεσες ενισχύσεις ως αντιστάθμισμα για τις ε, απολαβές ε, των γεωργών. Πολλοί τομεί βέβαια δεν συμφωνούν, αλλά αν εκείνοι δεν φρόντιζαν τα υπέροχα τοπία μας και δεν παρήγαγαν τρόφιμα, κρίμα θα ήταν. Συγγνώμη, αφήστε με, δύο σύντομε σύντομες παρατηρήσεις. Ε, ε, μιλάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία για την πείνα στον κόσμο, μάλιστα. Πρέπει να παράγουμε πολλά περισσότερα για να θρέψουμε τον πληθυσμό ολάκερης της γης. Οι Γεωργοί έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να συμβάλλουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλλει. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο να σκεφτόμαστε τα περί αγρανάπαυσης. Μία τελευταία παρατήρηση τώρα για το ανώτατο όριο. Θα το συζητήσουμε και πάλι βέβαια το θέμα. Συγγνώμη, μία, μία απαντησούλα θα δώσω στον κύριο Μποβέ. Αφήστε με. Όχι. Ευχαριστούμε κύριε Αλλούλη. Μα μία απαντησούλα γιατί επιτέθηκε στον ε, παλιό φίλο μου Μάνσχολτ. Ο κύριος Μπόβε δεν ξέρω αν είναι και πολύ νεότερος από μένα, αλλά ε, ε, συνέβαλε επίση ε, στην κατάρτιση τη κοινή γεωργική πολιτική στην εποχή του κυρίου Μάνσχολτ, όπω και εγώ, αλλά η πολιτική του κυρίου Μάνσχολτ εστέφθη με απόλυτη επιτυχία και η γεωργή τότε ήταν πολύ πιο αποδοτική από ό,τι είχε προβλέψει ο κύριο Μάνσχολτ. Συγγνώμη το λέω, γιατί έπρεπε να υπερασπιστώ το φίλο μου. Κάποιοι συνάδελφοι υπερέβησαν ε, τον ε, χρόνο, ζητώσαν από όσους δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Κύριε Επίτροπε, ήρθατε σήμερα εδώ και εκτεθήκατε ουσιαστικά σε ένα σωρό σχόλια από την αριστερά μέχρι τη δεξιά από τα έργα του Κοινοβουλίου. Θα σας ε, παρακαλέσουμε λοιπόν να αξιοποιήσετε την ισχύ του αξιώματός σας για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, ε, γιατί και εμείς αυτό θα το πράξουμε καθότι μας δίνεται η εξουσία από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σας δίνω τώρα το λόγο για να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δώσω κάποιες ε, πολύ γρήγορες απαντήσεις. Δυστυχώς ε, έχω και άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις και υπερβήκαμε κάπως το χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν με κάθε σεβασμό, αν μου επιτρέπετε, δεν θα επισέλθω σε αυτή τη φάση σε λεπτομέρειες επαναλαμβάνω, έχουμε και στοιχεία συγκεκριμένα, έχουμε λεπτομέρειες, δεν τα έχουμε αναλύσει ακόμα όμως αυτά τα και γι' αυτό δεν θεώρησα σκόπιμα να τα παρουσιάσω σε εσάς. Καταλαβαίνω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Παραδείγματο ότι αυτό που είπε η κυρία Ρέινιξ, ότι υπάρχει ένα, μια έκθεση από το έρχεται άλλη μια τώρα από την Κομισιόν η νομοθετική πρωτοβουλία ε, ε, είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής και η Επιτροπή θα παρουσιάσει ανακοίνωση και μετά ε, θα παρουσιάσει τα νομοθετήματα. Τις λεπτομέρειες που θέλετε θα τις βρείτε στα επικείμενα νομοθετήματα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Επίση, ήδη το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν τη δυνατότητα επί τη βάση των γενικών προσανατολισμών να υποβάλουν και άλλε προτάσει, όπω ε, η έκθεση του Κοινοβουλίου που προτείνει κάποιου προσανατολισμού. Απλούστευση και πράσινοποίηση σε εισαγωγικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίφαση. Συμφωνώ με αυτά που είπε. Ποιο το είπε, ο κύριο Φόλο, δεν θυμάμαι ακριβώ, ή ο κύριο Νταντά. Ε, πρασινοποίηση αν υπάρχει και, και απλούστευση της πολλαπλής συμμόρφωσης. Ναι, το κατάλαβα, το κατέγραψα. Αυτός είναι ο στόχος μου Η πολυπλοκότητα της υλοποίησης της κοινή γεωρικής πολιτικής ε, δεν έχει σχέση μόνο με τα νομοθετήματα των, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί η εκτέλεση, η υλοποίηση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη ορίζουν το νομικό πλαίσιο υλοποίησης. Ε, ε, μην το ξεχνάτε, γιατί τις τα τελευταία τρία έτη, αν κάποιο προέβησε σε απλούστευση, αυτή ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να έχουμε ε, συζητήσει. εσφαλμένες συζητήσεις. Χρειάζεται στόχευση. Κυρία Μαγκίνες, εγώ ε, δεν έρχομαι εδώ σε αμυντική στάση. Απλώ πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλοί αναρωτιούνται και εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο για το μέλλον της ε, κοινή ε, γεωργική πολιτική. Και μην ξεχνάτε ότι πρέπει να έχουμε μια επιχειρηματολογία που να πείθηκε τους έξω. Αυτό είναι μεταξύ άλλων ε, ο στόχος της ανακοίνωσης. Πρέπει να δράσουμε όμως τώρα, πριν είναι αργά. Δεν πρόκειται για αμυντική στάση, απλώς θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό και να ενεργήσουμε εγκαίρως, να το διευκρινίσουμε εγκαίρως. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συμφωνίες, το επανέλαβα, στόχος αυτής της μεταρρύθμισης δεν είναι είτε να ενισχύσετε να αποδυναμώσει τις διεθνείς συμφωνίες. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Η δική μου θέση ε, ξέρω ποια είναι και θα παίξω το διαπραγματευτικό μου χαρτί. Και μπορείτε να με κατηγορήσετε τα πάντα, αλλά όχι για έλλειψη διαφάνεια ε, απέναντι στο Κοινοβούλιο ή για έλλειψη σαφήνεια. Σε ό,τι αφορά είτε το γάλα, είτε τη ζάχαρη, είτε άλλου τομεί, ε, δεν μπορούν να υπάρξουν ε, τομεακή, δεν μπορούμε να κάνουμε, να μιλήσουμε για τομεακές ε, μεταρρυθμίσεις. Ε. Πρέπει να σεβαστούμε το ρόλο της ανακοίνωσης ε, και του εγγράφου συγκεκριμένου που είναι έγγραφο προσανατολισμού όπως είπα. Θα έχετε στη συνέχεια κάποια στοιχεία και για τη ζάχαρη θα γίνουν μεταρρυθμίσεις. Τώρα θα δούμε κατά πόσον θα τις διευκρινίσουμε στην συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ή στο πλαίσιο κάποιας άλλης μεταρρύθμισης. Στόχος μου πάντως δεν ήταν επί του παρόντος να ασχοληθώ Τώρα, πώς μπορούμε να ε, σχετίσουμε τα ειδικά θέματα ε, και με την ευελιξία. Όταν ζητούν τα κράτη-μέλη ευελιξία, εγώ του ζητώ από την πλευρά μου να τη χρησιμοποιήσουν για να τη δώσουν αξία αυτή τη ευελιξία. Εδώ μιλάμε για συμπληρωματικότητα ουσιαστικά μεταξύ ε, των γενικών στόχων που εξυπηρετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των ειδικότερων στόχων που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τις μειονεκτικές περιοχές, τα ειδικά μέτρα για τις μειονεκτικές περιοχές παραμένουν στο δεύτερο πυλώνα. Απλά στον πρώτο πυλώνα δεν υπάρχει ουσιαστικά ε, κατά ανάγκη μια μεταφορά, αλλά στον πρώτο πυλώνα, στο πλαίσιο αυτού του επανακαθορισμού των κριτηρίων διανομής, δίνουμε τη δυνατότητα να ληφθεί υπόψη με μια συμπληρωματική πληρωμή περιορισμένου ύψους που θα προσθεθεί στη βασική πληρωμή, να ληφθεί υπόψη ο της, ε, να ληφθούν υπόψη ουσιαστικά οι μειονεκτικές περιοχές. Φυσικά, υπάρχουν και συγκεκριμένες ειδικέ ε, πληρωμές χρηματοδοτήσεις από τα κράτη-μέλη για τις μειονεκτικές περιοχές, παραδείγματος χάρη για το κόστος μεταφοράς του γάλακτος ή άλλων προϊόντων κτλ. κτλ. Υπάρχουν ειδικά μέτρα και όλα αυτά παραμένουν εντός του δεύτερου πυλώνα. Σε ό,τι αφορά την αποσύνδεση πράγματι ε, το προτείνουμε το πώς ε, θα έλθει στη συνέχεια, πώς θα χρησιμοποιηθεί. Μάλλον η σύνδεση. Τώρα το θέμα είναι να προστεθεί στον πρώτο πυλόν η δυνατότητα να παραμείνει η σύνδεση, αλλά για κάποιου τομείς και για κάποιε συγκεκριμένε περιοχές εκεί έχουμε κάποιες αιτιολογίες. Το θέμα είναι να δώσουμε ένα μήνυμα και αυτό κάνουμε. Για τη δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων. Μεταβατική περίοδος. Είπα ε, και επαναλαμβάνω ότι νομίζω ότι χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος ε, που θα δούμε αν θα είναι λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη. Και θα δούμε τις ε, προτάσεις που θα έχουμε όταν προκάνουμε και εμείς τη δική μας πρόταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, επανέρχομαι. Καταλαβαίνω Καταλαβαίνω τι ανησυχίε πολλών από εσά για τον προπολογισμό. Είναι κάτι που με ανησυχεί και εμένα. Ο καλύτερο τρόπο να ανταποκριθούμε στην ανησυχία αυτή στο παρόν στάδιο είναι να κάνουμε μια συνεπή πρόταση για το μέλλον τη κοινή γεωργική πολιτική. Αλλά επαναλαμβάνω το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί έναν περιορισμένο προπολογισμό για πολύ σημαντικέ και παραδοσιακά κοινοτικέ πολιτικές και βέβαια πρέπει ταυτόχρονα να χρηματοδοτηθούν και νέε πολιτικέ. Κάτι που ζητούν από την Κομισιόν τα κράτη-μέλη αλλά και το Κοινοβούλιο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Εάν ζητούν από την Επιτροπή, ε, μάλλον λένε στην Επιτροπή ότι έχετε έναν ακόμα πιο περιορισμένο προπολογισμό, αλλά πρέπει να κάνετε περισσότερα πράγματα, η Κομισιόν πρέπει να βρει και αυτή κάποιε λύσει. Και μια από τι λύσει είναι να δει πώ θα εξισορροπήσει τι φιλοδοξίε ε, σε σχέση με τις διαφορετικές παραδοσιακές κοινοτικέ πολιτικές, να δούμε τι μέσα έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι, μέτρα σε ε, τι μέσα σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταλαβαίνω επίσης και βέβαια ταυτόχρονα είμαι και εγώ υπέρμαχος ενός σημαντικού γεωργικού προπολογισμού, αλλά ξέρω ότι πρέπει να κάνει και ο συνάδελφο Λεβαντόφσκι που έχει διάφορε επιλογέ να διαχειριστεί. Ελπίζω λοιπόν να μην βρεθούμε στην κατάσταση όπου θα πρέπει να θυσιάσουμε παραδοσιακέ πολιτικέ για να αντισταθμίσουμε άλλε πολιτικέ. Δεν είναι μόνο θέμα επιλογή μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών, αλλά είναι και θέμα επιλογή μεγέθου του συνολικού ευρωπαϊκού προπολογισμού. Δεν νομίζω τώρα ότι το έγγραφο ε, ανακοινώνει ή προβλέπει ουσιαστικά περισσότερη γραφειοκρατία. Η απλούστευση αφορά μόνο τον ευρωπαϊκό κανονισμό και θα το προσέξω πολύ, σας διαβεβαιώ. Ε, θα προσέξω να αποφύγω περι, περαιτέρω περιπλοκές. Δεν νομίζω ουσιαστικά ότι περιπλέκονται τα πράγματα ή ότι σε ό,τι αφορά τον έλεγχο επιτόπου, ότι υπάρχει κάτι πιο πολύπλοκο. Σε επίπεδο κρατών μελών είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, τροφική αλυσίδα, μου άρεσε αυτό που είπε η κυρία Μαγκίνες για την πράσινη γραφειοκρατία. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό οφείλεται στη δική μας ε, πρόταση για πρασίνισμα. Καλύτερη κατανομή και προσθέμενη αξία, είπα, σχετίζονται και με ζητήματα όπω είναι η διακύμανση. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτική γιατί υπερβαίνουν το γεωργικό τομέα όπω η αγροδιατροφική αλυσίδα που έχει να κάνει επίση με την πολιτική τη εσωτερική αγορά, με τη βιομηχανική πολιτική ή με την πολιτική ανταγωνισμού. Είναι ένα θέμα που το βλέπουμε και ξεχωριστά. Υπάρχει ένα φόρουμ για την γεωργοδιατροφική αλυσίδα το ξεκίνησε ο Επίτροπος Ταγιάννη με συνεργασία και με μένα και με τον κύριο Νταλή και με τον κύριο Μπαρνιέ. Επίσης έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε ένα σχέδιο προτάσεων και δράσεων για το θέμα αυτό και γιατί όχι θα μπορούσαμε ε, και στο πλαίσιο της Γκρι με, τον με τους κυρίους Μπαρνιέ, Γιάννη Νταλή να οργανώσουμε και μία ενημέρωση για να δείτε και εσείς περί τίνος πρόκειται. Κυρία μου λέτε ότι είναι πολύ ασαφή ο πρώτο πυλώνα και πολύ, πολλά, πράγματα περιέχει ο δεύτερος. Χαίρομαι που μου το λέτε αυτό, γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι ο δεύτερος πυλώνα δεν ήταν και τόσο γεμάτο, αλλά ότι ήταν πολύ γεμάτο ο πρώτος πυλώνα. Γιατί και εκεί λέμε στον πρώτο πυλώνα τι είδου άμεσε πληρωμέ, σε ποια κατηγορία. Μιλάμε για μικρέ γεωργικέ εκμεταλλεύσει μιλάμε για σύνδεση κτλ. Υπάρχουν πολλά ε, σε σχέση με τις άμεσες πληρώμες στον πρώτο πυλώνα. Τώρα, αν εσείς περιμένετε συγκεκριμένα κριτήρια διανομής, αυτό ή κατανομής, αυτός ε, είναι ο ρόλος του νομοθετικού πακέτου. Αυτό το πακέτο θα έχει αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια και εγώ δεν μπορώ τώρα να αναφέρω κάτι χωρί να γίνουν, όπω είπα και πριν, μελέτε επιπτώσεων πρώτα. Ο ε, κύριε Πατράου μου έκανε πάρα πολλέ ερωτήσει ε, που είναι πάρα πολύ λεπτομεριακέ και δεν μπορώ επομένω να απαντήσω τώρα. Αυτό το οποίο μπορώ να πω πάντω σε σχέση με τι Αζόρε και σε σχέση με τι ε, μειονεκτικέ περιοχέ και το επαναλαμβάνω ουσιαστικά είναι ότι έχουμε ένα μέσο το οποίο σκέφτομαι να το διατηρήσω και θέλω και να το μεταρρυθμίσουμε αν είναι δυνατόν για να μπορεί να τα αποκριθεί καλύτερα. Και θα έχουμε μια πρόταση μεταρρύθμισης αναδιάρθρωσης ε, υπό την καλή έννοια προς σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τις άκρως απόμακρες περιφέρειες και αυτές αποφελούνται στο πλαίσιο του δεύτερου πυλών από προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και θα έρθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις ε, για να ανταποκριθούμε ιδίως στο ζήτημα της διαφοροποίησης στις περιοχές αυτές. Σε ό,τι αφορά τώρα τα γαλακτοκομικά, αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε όταν ε, μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον τομέα του γάλακτος. Για την κυρία Γιούσο, η οποία μου λέει ότι ε, πράγματι, αν διαβάσετε το κείμενο θα δείτε ότι υπάρχουν αναφορές για αυτά που είπατε. Υπάρχει αναφορά στην επανεξισορρόπηση. Υπάρχουν απαντήσεις για τις ε, περιπτώσεις ε, έκτακτης ανάγκης, για καταστάσεις κρίσης. Υπάρχουν απαντήσεις για την παραγωγική γεωργία στο σκέλος της αγροτικής ανάπτυξης. Εγώ νομίζω ότι αντιθέτως με αυτό που είπατε υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Το αυτό το είπα. Αυτά είχα να πω. Σα ευχαριστώ πολύ. Ζητώ για μια ακόμη φορά, συγγνώμη αν δεν μπόρεσα να σα δώσω περισσότερε λεπτομέρειε στι απαντήσει μου, αλλά έχουμε την... θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συγκεκριμένο μπορώ. Παναλαμβάνω όμω αυτό που είπα και παλαιότερα στο Κοινοβούλιο. Α προσπαθήσουμε να μην χάσουμε το ε, δάσος ε, το δέντρο μόνο. Θα έρθουν και οι λεπτομέρειε. Παρακαλώ τους συντονιστές να με ακολουθήσουν στην κεκλεισμένα των θυρών συνεδρίωση που θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Πελίε τη